Good afternoon everyone. Καλό απόγευμα σε όλους. Παρακαλώ πάρτε θέσεις για να αρχίσουμε την δημόσια ακρόαση τη σημερινή. Καλώς ήρθατε στη δημόσια ακρόαση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την απαγόρευση της γλυφοσάτης και την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά ζανιοκτώνα. Αυτή η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών συνέλεξε πάνω από ένα εκατομμύριο, από ένα εκατομμύριο υπογραφές από πολλά και διάφορα κράτη-μέλη. Είναι τέταρτη επιτυχής πρωτοβουλία πολιτών από τη θέση ισχύ της Δίκης Λισαβόνας. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των χαίρεται ιδιαίτερα που ανέλαβε να οργανώσει αυτή την ε, δημόσια ακρόαση σε συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών, την Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Ο στόχος της σημερινής ακρόασης είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους οργανωτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ε, να παρουσιάσουν δημόσια εδώ σε μια πλατφόρμα, σε ένα φόρουμ την πρωτοβουλία τους και να ε, έχουν ένα επικοδομητικό διάλογο με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαιρόμαστε που ο Επίτροπος Αντριουκάητης, ε, ο Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δέχθηκε να παραστεί σήμερα εδώ και να συνεισφέρει στην συζήτηση μεταξύ των οργανωτών της πρωτοβουλίας και των μελών του Κοινοβουλίου. Ο στόχος είναι να απαγορευτεί η γλυφοσάτη, να αλλάξει η διαδικασία για την αξιολόγηση της γλυφοσάτης σε επιστημονικό επίπεδο και η εισαγωγή υποχρεωτικών στόχων μείωσης ό,τι αφορά τη χρήση νεοκτώνων. Όπω ξέρετε, το Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί πολλάκις με το θέμα αυτό. Τον Οκτώβριο στις 24 δεν συμφωνήσαμε με το σχέδιο νομοθετικής πράξης της Κομισιόν που πρότεινε την παράταση της, της άδειας για τη Λιφοσάτη για 10 χρόνια ε, κάποιες ε, προτάσεις που έχουν να κάνουν με την σταδιακή απομάκρυνση της γλυφοσάτης το 2022, αλλά αυτά δεν έγιναν αποδεκτά. Είχαμε μια συνάντηση και με την Επιτροπή Γεωργίας, μια κοινή δημόσια ακρόαση για τα πιο σημαντικά στοιχεία που αφορούν την γλυφοσάτη υπήρξαν, συμμετείχαν ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονε ε, των αρχών πιστοποίηση, συζητήθηκε η επιστημονική βάση για την αξιολόγηση κινδύνου τη γλυφοσάτη και ο, το, το πώ έχει αντιδράσει ο κλάδο τη ΗΠΑ στο πλαίσιο τη αξιολόγηση αυτή. Να πω δύο λόγια για τη δομή τη σημερινή συνάντηση. Στη, στην αρχή θα έχουμε μια παρουσίαση ε, τη ε, πρωτοβουλίας ε, πολιτών Στη συνέχεια θα μιλήσει ο κ. Ανδρουκάητης και ο κύριος Adrian Burns από την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών. Στη συνέχεια θα έχουμε τρεις γύρους συζητήσεων. Κάθε γύρο θα αφορά έναν από τους στόχους της πρωτοβουλίας πολιτών. Δηλαδή η απαγόρευση της γλυφωσάτης, δεύτερον η αλλαγή οι αλλαγέ στην διαδικασία επιστημονική αξιολόγηση των συνεκτώνα και τρίτον η πανευρωπαϊκή υποχρεωτικοί στόχοι για τη μείωση χρήσης ζωνιωτών. Και για του τρεις αυτούς ε, γύρους θα σας πω πώς θα προχωρήσουμε όταν φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, δεσποινίδα Μίκα Λεάντρο που εκπροσωπεί την Επιτροπή Πολιτών. Για 10 λεπτά παρακαλώ. Bonjour. Good afternoon. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους παριστάμενους στην αίθουσα αλλά και στους πολίτες που παρακολουθούν την ακρόαση μέσω του διαδικτύου. Καλησπέρα. Μίκλη Άντριου με λένε και εκπροσωπώ την Επιτροπή ε, των Πολιτών για αυτή την πρωτοβουλία πολιτών και εκπροσωπώ ε, αυτή, αυτό το φορέα. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Ευρωκοινοβούλιο και κυρίως της, ε, την Επιτροπή Περιβάλλοντος Γεωργίας, Βιομηχανίας και Αναφορών που μα προσεκάλεσαν να παρουσιάσουμε την πρωτοβουλία μα, η απαγόρευση τη γλυφωσάτης να προστατεύσουμε τον κόσμο και το περιβάλλον από τα τοξικά παρασυντοχτών ενός στόχος μας. Επίση, θα ήθελα να ξεκινήσω παραδεχόμενο ότι η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου πρόσφατα ψήφισε ψήφισμα που ζητά απαγόρευση τη γλυφωσάτης μέχρι το 2022. Αυτό αποδεικνύει πόσο σοβαρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη ανησυχίε των πολιτών. Όμω οι Ευρωπαίοι πολίτε υπήρξαν σαφεί. Θέλουν απαγόρευση και δεν θέλουμε να αναθεί η χρήση της γλυφοσάτης μέχρι τώρα. Η αρχή της πρόληψης θα πρέπει να εφαρμοστεί και η γλυφοσάτη θα πρέπει να αφαιρεθεί από τα διάφορα αγροτικά συστήματα. Λοιπόν, το πρωτοβουλία μα ζητά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει στα κράτη-μέλη μια απαγόρευση για την γλυφοσάτη. Να μεταρρυθμιστεί η διαδικασία έγκριση παρασιτοκτόνων και καθορίσουν υποχρεωτική στόχη μειώσεω τη χρήση παρασιτοκτόνων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνάδελφοί μου εδώ θα παρουσιάσουν καθέναν από του στόχου λεπτομερώ. Εγώ θα ξεκινήσω ακροθυγώ περιγράφοντα την όλη δομή τη πρωτοβουλία των πολιτών συγκεκριμένη. Καταρχά, πρώτο στόχο είναι προφανώ η απαγόρευση τη γλυφωσάτη. Γιατί? Διότι υπάρχει συνένεση επιστημονική ότι είναι τοξική ουσία. Και οι ρυθμιστικοί φορεί τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω συμφωνούν με αυτό. Αυτό από μόνο του πρέπει να αρκεί για να είμαστε προσεκτικοί. Επιπλέον, διεθνεί φορεί πασίγνωστοι για την έρευνα του τον και οι διάφοροι φορείς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχουν καθορίσει ότι είναι ε, πιθανός και καρκινογόνος ουσία η γλυφοσάτη. Η, τοξικότητα και οι καρκινογόνε καρκινογόνες ε, επιρροές της γλυφοσάτη βρίσκονται παντού. Ε, βρίσκομαι σε κατάλοιπα πολλών βασικών τροφίμων όπως είναι το ψωμί και τα διάφορα τρόφιμα για τα μωρά και σε διάφορα στοιχεία που βρίσκουμε στον οργανισμό μας. Ε, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι που κάνουν δοκιμασίε ούρων ε, για γλυφοσάτη μπορεί να αναμένουν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την παρουσία γλυφοσάτη στα ούρα του. Επιπλέον, είναι ένα παρασιτοκτόνο που έχει οδηγήσει σε επιδείνωση των οικοσυστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σημαντική αρνητική επιρροή στην βιοπικιλότητα. Κάτι που το δέχονται ρυθμιστικοί φορεί τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Επόμενο, τώρα θέλουμε πλήρη μεταρρύθμιση της διαδικασία αδειοδότηση των παρασιτοκτόνων και αυτό είναι ο δεύτερος στόχος. Γιατί, διότι η γλυφοσάτη είναι ένα σύμβολο για όλα όσα είναι λανθασμένο όσον αφορά στι φυσικές διαδικασίε. Γι' αυτό επίση ζητούμε μεταρρύθμιση των σχετικών διαδικασιών, να εξασφαλίσουμε ότι η αξιολόγηση και η διαδικασία είναι αντικειμενικά διαφανή ε, και ανεξάρτητα ω προσεγγίσει, όπω απαιτείται από την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση των Παρασιτοκτών. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτό που συμβαίνει με γλυφοσάτη έχει συμβεί και με άλλα παρασιτοκτών στο παρελθόν και θα συμβεί και ξανά αν δεν δραστηριοποιηθούμε για αλλαγή του συστήματο. Ε, Τέλο. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει υποχρεωτικού στόχου μειώσεω για τη χρήση παρασιτοκτών ω μέλη. Θα πρέπει να πάμε σε ένα μέλλον χωρί παρασιτοκτόνα. Να περιγράψω γιατί αυτό ο στόχο είναι σημαντικό για μα. Σήμερα έχουμε οδηγία για βιώσιμη χρήση των παρασιτοκτόνων. Ένα παρασιτοκτόνο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν όσοι άλλε μέθοδοι δεν μπορούν να έχουν αποτελέσματα και δίνει εντολή στα κράτη μέσα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να θεσπίσουν συγκεκριμένου στόχου και μέτρα για τη μείωση τη χρήση παρασιτοκτόνων αλλά δυστυχώς τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν επαρκώς την οδηγία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα δεν έχει αξιολογήσει τις συνέπειες της οδηγίας και της μη σωστής εφαρμογής. Η οδηγία θα πρέπει να ενισχυθεί. Θα πρέπει να βάζουμε στόχους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσης, θα πρέπει να οδεύονται από μέτρα υποστήριξη του γεωργούς, ούτως ώστε αποτελεσματικά να μειωθεί η χρήση των παρασιτοκτόνων. Αυτό είναι σημαντικό, διότι πέραν από την γλυφοσάτη, πάνω από 500 άλλα παρασιτοκτόνα ε, έχουν αδειοδοτηθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν τα τοξικά παρασιτοκτόνα αποσυρθούν από την αγορά ή περιοριστεί χρήση αυτών, η μηχανία η των παρασιτοκτόνων αντικαθιστά αυτέ τι ουσίε με άλλε χημικέ ουσίε και πολύ γρήγορα μάλιστα. Και η τα χημικά που χρησιμοποιείται στα παρασιτοκτόνα μπορεί να επηρεάσουν του οργανισμού και το περιβάλλον στο οποίο ζουν και από το οποίο εξαρτώνται. Και ενδεχομένω θα έχουμε σοβαρέ οικολογικέ συνέπειε. Τέλο, ουσιαστικά τα οικοσυστήματα κινδυνεύουν η γονιμότητα του εδάφους, η γονιμοποίηση των φυτών και παραδόξως διάφορες φυσικές διαδικασίες για τον έλεγχο των παρασίτων. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική στόχη. 1,3 εκατομμύρια πολίτες υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών έχει τύχει υποστηρίξεως σε ένα πεντάμινο. Λιγότερο από πέντε μήνες. Αυτό δεν είχε επιτευχθεί ποτέ πριν. Είναι ένα πραγματικό ρεκόρ ε, κατέστη εφικτό αυτό χάρη σε μια συμμαχία απίστευτη. Πάνω από 100 οργανώσει των κοινωνία των πολιτών, από συνδικάτα, ενώσεις ε, γεωργών, ομάδες θυμάτων, ΜΚΟ, προστασία του περιβάλλοντος και πολλοί άλλοι φορεί συνεργάστηκαν και όχι μόνο αυτοί. Στο επίκεντρο αυτή της πρωτοβουλίας των πολιτών είναι οι ίδιοι οι πολίτες ήταν ο βασικό οδηγό, η κινητήρια δύναμη. Δεν θα ήταν δυνατόν χωρί να συμμετάσχουν οι πολίτε να το πετύχουμε αυτό. Πάνω από 250.000 υπογραφέ συνελέγησαν έξω από σχολεία, μαγαζιά, σε πάρκα, από πολίτε στι γειτονιέ του, στι πόλει του και στην Ήπεθρο, σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, για μια στιγμή να σα δείξω και κάποιε εικόνε από την συλλογή των υπογραφών. Έχω κάποιε εικόνε να σας δείξω. Όπως βλέπετε έγινε πολλή δουλειά. Η επιτυχία δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν δράση. Κυρίως όσον αφορά την γλυφοσάτη και γενικότερα για τα παρασιτοκτόνα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν θέσει την εμπιστοσύνη τους στα χέρια των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και στο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πάει στα σοβαρά. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν και οι ανησυχίες μας είναι θεμητές το ευρωπαϊκό κοινό μίλησε μέσω του Κοινοβουλίου, μέσω της Ευρωπαϊκής Πολι... ε, Πρωτοβουλίας Πολιτών και από διάφορες δημοσκοπήσεις και έχουν δείξει ότι η μεγάλη πλειοψηφία θέλει την απαγόρευση της γλυφωσάτης. Η θέσπιση νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα της σωστή δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η διαδικασία διαμόρφωσης πολιτική όσον αφορά την γλυφωσάτη δεν έχει ανταποκριθεί στα πρότυπα από το καλοκαίρι του 2016 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκτηνε την αδειοδότηση για αυτό το αμφίσιμο προϊόν χωρίς ειδική πλειοψηφία ε, έκαναν προρία, προσπάθεια να εισακουστεί φωνή τους οι πολίτες, να ακουστεί μέχρι τους διαδρόμους ε, της εξουσίας της Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες προσπάθησαν να προωθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τότε, από το καλοκαίρι και απευθύνουμε έκκληση στο ύψιστο δυνατό επίπεδο μέσω τη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλίας Πολιτών. Όμως, παρά τις επιτυχίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν άλλαξε την προσέγγιση της αφορά το θέμα αυτό, ούτε προσπάθησε να βρει μια αποδεκτή λύση. Ε, τα κράτη-μέλη συνεχώ λένε όχι στην γλυφωσάτη, όλο και περισσότερε χώρε λένε όχι στην γλυφωσάτη και έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά να ηγηθεί και να προτείνει μια απαγόρευση. Να μην ανανεωθεί η χρήση τη γλυφωσάτη. Αυτό ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Οι πολιτικές αποφάσεις όπως αυτή για τη Γλυφωσάτη απαιτούν την ηγεσία ανθρώπων με όραμα, εκείνων που θέλουν να σταθούν και να προστατεύσουν τους απλούς Ευρωπαίους πολίτες κατά των χρημάτων, της εξουσίας και των απειλών των πολυεθνικών εταιριών. Η Ευρώπη απελπιστικά χρειάζεται οραματιστές όπως αυτούς για να ξεφύγουμε από την εθισμό μας στα χημικά και προς ένα μέλλον χωρίς παρασιτοκτόνα. Δεν διατηνόμεθα ότι θα είναι κάτι ανώδυνο να αλλαγούμε από αυτή τη συνέχεια, από τον εθισμό, τα παρασυτοκτόνα και τα χημικά. Χρειάζεται συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω, σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη. Εξασφαλίσουμε ότι οι γεωργοί θα τύχουν και ε, υποστήριξη στην απαγόρευση και να βρεθούν βιώσιμε εναλλακτικέ λύσει που χρησιμοποιούνται και να είναι προσβάσιμε για του γεωργού. Αλλά το κλειδί είναι ότι λύσει υπάρχουν. Υπάρχουν Ευρωπαίοι γεωργοί που ήδη καλλιεργούν χωρί να χρησιμοποιούν γλυφοσάτη και δεν χρησιμοποιούν καν παρασιτοκτόνα. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε μακριά από ένα μέλλον χωρίς παρασιτοκτόνα, στο βαθμό που διατηρείται η πολιτική βούληση για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους. Το 2009 η Ευρώπη αποφάσισε να θετήσει την πιο προστατευτική νομοθεσία τα παρασιτοκτόνα στον κόσμο. Με βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών. Είναι λοιπόν νόμιμο και θεμητό οι πολίτε να αναμένουν τέτοιε διατάξει αυτή τη πρότυπη νομοθεσία πραγματικά ότι θα εφαρμοστούν και θα χρησιμοποιηθούν. Κάτι που δεν ισχύει τώρα. Η περίπτωση τη γλυφωσάτη δείχνει καταφανώ ότι οι δύο σημαντικέ βελτιώσει τη νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ενώση για τα Πασιτοκτόνα δεν εφαρμόζονται από τι αρμόδιε αρχέ. Η προσέγγιση βάσει των κινδύνων και ανεξάρτητη αξιολόγηση μέσω τη επιστημονική τεκμηρίωση η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την κατεύθυνσή της όσον αφορά τα παρασιτοκτόνα. Αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών να υπηρετήσει σαν, ένα, σαν κόδωνα συναγερμού για να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι υπεύθυνη πρωτίστως για τους πολίτες της και όχι για τις ε, πολυεθνικές εταιρείε. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια επιλογή σήμερα. Έχει πραγματική δυνατότητα να ηγηθεί όσον αφορά τη βιώσιμη γεωργία του μέλλοντος χωρίς ε, τοξικά παρασιτοκτόνα. Θα ήθελα να κλείσω με μια σύντομη παράθεση ενός Γάλλου πολίτου. Είπε, Ήδη άλλαξαμε. Η Μιριέλ Παπέ. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε. Κάθε δισταγμό και αναβολή αποφάσει έχει ε, ε, συνέπειε για την υγεία και το περιβάλλον. Πρέπει να λάβουμε μια θαραλέα σήμερα απόφαση. Και αυτή είναι μια υπέροχη ευκαιρία, ούτω ώστε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να, α, να δείξουν σωστή εικόνα έναντι των πολιτών που ταλαιπωρούνται οικονομικά. Και από άλλους. Λοιπόν, καλούνται οι πολίτε, καλούν οι πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν το σωστό. Και αυτή είναι η ευκαιρία σα να το δοκιμάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος, ο κ. Ανδρουκάητης έχει το λόγο. Για ένα πεντάλεπτο. Ε, ε, αξιότιμη Πρόεδρε της Επιτροπής, ε, αξιότιμη Αντιπρόεδρε της Επιτροπής Αναφορών. Καλώς ε, σας βρήκα. Σήμερα η συνάντησή μας αποτελεί μια επίσημη συνάντηση ε, για την ε, συζήτηση της πρωτοβουλίας των πολιτών που ονομάζεται «Απαγόρευση της γλυφοσάτης» και θα υπάρξει και μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας όπως έγινε και τον περασμένο μήνα στις 23 ε, Οκτωβρίου στην Κομισιόν. Σήμερα έχουμε ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων την συμμετοχή μελών από την πρωτοβουλία και από τις σχετιζόμενες επιτροπές, τις επιτροπές ΠΕΤΗ, ΉΤΡΕ και ΆΓΡΙ και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους ε, διοργανωτές αυτής της πρωτοβουλίας ε, που πραγματικά ε, ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχει η συνθήκη της Λισαβόνης, Λισαβόνας και θέτουν ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι μια τέτοια συμμετοχή μπορεί να οδηγήσει στην αμοιβαία κατανόηση ευαίσθητων θεμάτων και να έχουμε μια καλύτερη συνεισφορά στον ορισμό των μελλοντικών θεμάτων. Έτσι η Κομισιόν καλωσορίζει την κινητοποίηση των πολιτών για το θέμα των ε, φυτοφαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ε, αυτά τα ζητήματα δεν περιορίζονται σε μία απλή απόφαση, αλλά θέτουν γενικότερα θέματα σχετικά με την ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παρασιτοκτόνα, τα οποία ποτέ δεν ήταν σε διαγωνισμό μορφιάς και ποτέ δεν θα, ήταν και, ε, δεν θα είναι και στο νούμερο ένα της δημοφιλίας μεταξύ των πολιτών. Όμως ε, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκής ε, τροφή, ότι οι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά ή να καταστρέψουν τα ζυζάνια που βλάπτουν ε, την ε, ε, σοδιά τους. Ας πούμε, στο παρελθόν, όταν είχαμε τα προβλήματα με την πατάτα στην Ιρλανδία, αν υπήρχαν αυτά τα ζυζανιοκτώνα θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Θυμάστε την ιστορία. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ασθένειες που χρειάζονται τακτικά προστατευτικά μέτρα. Παρ' όλα αυτά η παραγωγή των τροφών, των τροφίμων και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένα και θα πρέπει να υπάρξει μία ε, συνεχής παρακολούθηση και η κοινωνία να μεταστραφεί προς μία πιο πράσινη και βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Στην κοινή γεωργική πολιτική έχουμε την προώθηση της ε, ε, βιολογικής γεωργίας, ένα σύστημα συμβουλευτικής ε, μέτρα ε, για την ε, αγροτική ανάπτυξη, το πρασίνισμα της οικονομίας και πολλά άλλα ερευνητικά project. Αν θέλουμε λοιπόν να πάμε σε μια πιο ανθεκτική και πιο ηθική παραγωγή τροφίμων που θα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του μέλλοντος, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο όλα τα ε, διαθέσιμα εργαλεία. Θεωρώ ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των παρασύτων θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι οποιοδήποτε μελλοντικού συστήματος παραγωγής τροφίμων. Όσον αφορά στο περιεχόμενο της πρωτοβουλίας, να διασαφηνίσω ότι η Κομισιόν δεν είναι ο μόνος παράγοντας ε, που εμπλέκεται στο σύστημα το ρυθμιστικό που διέπει την έγκριση των παρασιτοκτόνων και τα κράτη-μέλη παίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση, την έγκριση και την αδειοδότηση και γι' αυτό θα, θα πρέπει να θεωρούνται ισότιμοι εταίροι στο σύστημα έγκρισης και αδειοδότησης. Ε, πρώτον λοιπόν έχουμε την έγκριση της ε, δραστικής ουσίας, ε, μετά έχουμε την αδειοδότηση του προϊόντος που την περιέχει στα κράτη-μέλη και όλα αυτά βασίζονται στην αρχή της επικουρικότητας. Αυτό δείχνει επίσης και τις διαφορές στις κλιματικές, αργονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες στα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν η πρωτοβουλία των πολιτών δεν πρέπει να απευθύνεται μόνο στην Κομισιόν αλλά και στα κράτη-μέλη τα οποία έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες ε, σε συνδυασμό με αυτές τις Κομισιόν. Πριν κλείσω να θέσω ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τελικά όλοι θέλουν το ίδιο αποτέλεσμα. Όλοι μας πασχίζουμε για τον ίδιο σκοπό. Ασφαλή τροφή που παράγεται με ηθικό και βιώσιμο αλλά και φιλικό προς το περιβάλλον ε, τρόπο με τις ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία μας. Είναι κοινή λογική. Η συνεργασία όλων των εταίρων για την προστασία των, ε, της υγείας και των πολιτών είναι μια κοινωνική ευθύνη που έχουμε και εμείς και την οφείλουμε σε εμά και στις μελλοντικέ γενές. Ο στόχος μας παραμένει λοιπόν πρώτα να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των παρασιτοκτόνων, δεύτερον να ε, ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους και να προσπαθήσουμε να βρούμε λιγότερο βλαπτικές και επιθετικές εναλλακτικές. Η Κομισιόν έχει ε, αναλάβει στεναρή δράση όλα αυτά τα χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση και ε, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα προϊόντα. Η οδηγία για τη χρήση των παρασιτοκτόνων μας δίνει τη δυνατότητα να μειώσουμε τους κινδύνους που προέρχονται από την κακή χρήση ή την υπερβολική χρήση των ε, παρασιτοκτόνων. Είναι η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν ένα σωστό τρόπο ε, να το επιδιώξουμε. Η Κομισιόν έχει ξεκαθαρίσει ότι χρειάζεται πρόοδο από την πλευρά των κρατών μελών. Η έκθεσή μα δείχνει ότι η εφαρμογή τη οδηγία στα κράτη-μέλη δεν είναι η ίδια ε, μπορούν να κάνουν περισσότερα τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται δημόσια ενημέρωση και να υπάρχει ελάχιστη χρήση σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα πάρκα, κοντά στα σχολεία κτλ. Επίσης θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις ε, καλύτερες τεχνικές, ολοκληρωμένες τεχνικές διαχείρισης ε, των ε, παρασιτοκτόνων. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε κράτος μέλος. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και αδειμονώ για μια γεμάτη πληροφορίες και επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα πρόεδρο τη Επιτροπή Γεωργία και Περιβάλλοντο τη Επιτροπή των Περίπτωσεων Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ο κ. Μπέρντ, έχει το λόγο δημιουργήθηκε με τη συνθήκη της Ρώμης. Ε, αποτελείται από τους εκπρόσωπους των εργοδοτών, των εργαζομένων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σε αυτό το τμήμα ε, συμμετέχουν οι εμπειρογνώμονες προσθέσεις ομάδες που ασχολούνται με το, τη γεωργία, την ε, γεωργική ανάπτυξη και το περιβάλλον. Να πω ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμη και σημαντική αυτή η διαδικασία της πρωτοβουλίας των πολιτών. Αυτό επιτρέπει μια επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Καλωσορίζουμε λοιπόν την πρόσθεση της Κομισιόν ε, για απλοποίηση αυτών των διαδικασιών. Προετοιμάζουμε μάλιστα σχετική γνωμοδότηση. Εμείς είμαστε μια γέφυρα μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης ε, και, της, ε, και των θεσμών της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να μπορούν να συζητούνται οι πρωτοβουλίες αυτές στα θεσμικά όργανα. έχουμε οργανώσει μία συζήτηση με όλους τους εμπλεκομένους φορεί στη δική μας επιτροπή και μπόρεσαν ε, οι εκπρόσωποι της πρωτοβουλία των πολιτών να παρουσιάσουν ε, την υπόθεση αυτή, το, τα επιχειρήματά τους στην ολομέλειά μας ε, με 450 μέλη. Και τα θέματα αυτά συζητήθηκαν ενδελεχώς. Δεν υπήρξε, δεν υπήρξε συνένεση μεταξύ των εκπροσώπων της Κοινωνίας των πολιτών για το κατά πόσο ε, θα πρέπει να απαγορευτεί η γλυφοσάτη. Οι αρχικές συζητήσεις απέδειξαν ότι υπάρχει απόκληση απόψεων. Βεβαίως η πρωτοβουλία αυτή ε, των πολιτών είναι καθρέφτης κοινωνίας, οπότε δεν θα εκπλαγείτε που σας το λέω αυτό. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω ε, την θέση, τις θέσεις που ακούστηκαν. Κανείς δεν θέλει βεβαίως ε, χημικά προϊόντα τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία στο περιβάλλον και στα τρόφιμα. Ε, και βεβαίω οι πολιτικοί δίνοντε βρίσκονται σε δύσκολη θέση, διότι διάφορε ακαδημαϊκές μελέτες οδηγούν σε αντιφατικά συμπεράσματα. Τέλος, ε, έχουν εκφράστηκαν ανησυχίες ε, για το γεγονός ότι κάποιες πολυεθνικέ έχουν τεράστια εξουσία, αλλά και κάποιες περιβαλλοντικές ομάδες, για να προωθήσουν θέσει που δεν είναι επωφελείς για τη συζήτηση αυτή. Μια συζήτηση πρέπει να βασίζεται ε, σε γεγονότα, σε δεδομένα και όχι σε ε, παραπληροφόρηση. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δώσετε να παρουσιάσουμε αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από την Επιτροπή ε, Αναφορών για τρία λεπτά ο κύριος Τσάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Επιτροπής των Αναφορών ε, της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμείς ε, χαιρόμαστε που μπορεί να λάβει, μπορεί χώρα αυτή η συζήτηση για την πρωτοβουλία πολιτών, για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Ω αντιπρόεδρο τη επιτροπή Αναφορών, χαίρομαι ιδιαίτερα που άλλη μία πρωτοβουλία πολιτών φτάνει έω εδώ σε μια δημόσια ακρόαση στο Κοινοβούλιο. Όπω έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια του κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών, δεν είναι εύκολο πάντα για του πολιτέ να φτάσουν σε αυτό το στάδιο να μπορέσουν να συλλέξουν ένα εκατομμύριο υπογραφές που χρειάζονται. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το νομικό πλαίσιο της Επιτροπής Αναφορών, το, το νομικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας μάλλον πολιτών, ε, βρίσκεται υπό αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε πάρει θέση ακόμα για τη νέα νομοθετική πρόταση της Κομισιόν έτσι ώστε αυτή η πρωτοβουλία να είναι πιο φιλική προς τους πολίτες και να είναι ένα πιο προσβάσιμο εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας. Τέλος, να πω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι έχουμε λάβει πολλές αναφορές από αυτού του ζητήματος για απαγόρευση και περιορισμό της χρήσης γλυφοσάτης που δείχνει, κάτι που δείχνει ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για πολλούς συμπολίτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτούς τους λόγους εμείς καλωσορίζουμε αυτή την ακρόαση ως μια ευκαιρία να εμβαθυνθεί αυτή η συζήτηση και να βρούμε λύσεις ε, που να προσανατολίζονται προς ε, το όφελος των συμπολιτών μας. Εύχομαι λοιπόν να έχουμε σήμερα έναν πολύ επικοδομητικό διάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τις αρχικές παρεμβάσεις και όπως είπαν νωρίτερα, τώρα θα περάσουμε στην εξέταση του κάθε στόχου της πρωτοβουλίας ξεχωριστά. Και θα ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση του πρώτου στόχου από την ε, Επιτροπή ε, της Πρωτοβουλίας Πολιτών. Στη συνέχεια θα έχουμε ερωτήσεις από τα μέλη του Κοινοβουλίου και τα συμπεράσματα. Αυτή θα είναι η δομή και για, την κάθε, ε, για τον κάθε στόχο. Δύο λεπτά παρακαλώ όμως ε, στις ερωτήσεις εννοώ των Ευρωβουλευτών. Πρώτα, πρώτος στόχος, απαγόρευση της κλειφωσάτης. Θα καλέσουμε λοιπόν τη Φραντσίσκα Αχτερμπεργκ, εκπρόσωπο της Επιτροπής Πολιτών για να μας παρουσιάσει για πέντε λεπτά αυτόν τον στόχο. Παρακαλώ. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που μας υποδεχθήκατε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Oh, oh, Α, αυτό είναι το μικρόφωνο μου, ωραία, πιο εύκολα έτσι. Θα ήθελα λοιπόν να περιμένω τη διαφάνεια πρώτα. Να παρουσιάσω τον πρώτο στόχο. Πρέπει να ζητήσουμε και τη βοήθεια της τεχνικής ομάδας, λοιπόν. Εν τω μεταξύ με την ευκαιρία να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο εκ για την πολύ επίκαιρη διοργάνωση της ακροάσεως. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουν δυνατότητα ήδη τώρα πριν τη λήψη τελικής αποφάσεως επί γλυφωσάτης να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, απαγόρευση της γλυφωσάτης, με τα χαρά σε επαναλαμβάνω τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες ζητούν αυτή την απαγόρευση Καταρχάς η γλυφοσάτη δημιουργεί καταστροφικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα και σχεδιαστεί να σκοτώνει τα φυτά αδιακρίτως, κάθε είδους φυτό. Επίσης είναι τοξική ουσία που επηρεάζει και άλλα είδη που δεν είναι φυτά. Ε, όπως είναι αράχνες, ερπετά και διάφοροι άλλοι οργανισμοί καταστρέφονται παρόλο που είναι ευεργετικοί οργανισμοί. Η τοξικότητα της γλυφοσάτης μαζί με τις άλλες συνέπειες που έχει χρήση στο περιβάλλον καθιστά αυτή την ουσία μία μηχανή που σκοτώνει, μηχανή δολοφόνο. Το ίδιο έτσι του παρουσιάζουν την ουσία και η ίδια παραγωγή της ουσίας. δεύτερον, η γλυφοσάτη επίσης ε, είναι σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Έχει ταξινομηθεί σαν πιθανότατο αίτιο ε, για καρκίνο από τον οργανισμό, από την υπηρεσία για τον καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και έχει πολλά άλλα αρνητικά αποτελέσματα όπως σεξουαλική ανάπτυξη, αναπαραγωγικότητα, νευροτοξικότητα. Έχει όλες αυτές οι συνέπειες αρνητικές. Τώρα, η νομοθεσία για τα παρασιτοκτόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι τα παρασιτοκτόνα που είναι εγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να έχουν απαράδεκτο αντίκτυπο για το περιβάλλον, ούτε επιβλαβή συνέπεια για την ανθρώπινη υγεία συμπεριλαμβανομένης και της υγείας όλων των ευάλωτων ε, πληθυσμών. Αυτό σημαίνει όλος ιδιαίτερος ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ουσίες που είναι καρκινογόνες σύμφωνα με τα κριτήρια του ΆΙΑΚ, της Υπηρεσίας του Οργανισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον καρκίνο. Οι αξιολογήσεις της ΕΦΣΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν μεγάλους κινδύνους μακροπροθεσμού για τα θηλαστικά και τα πτηνά με κάποια κενά στον αυτά τα στοιχεία, οπότε ο υψηλό κινδύνο δεν έχει αποδειχτεί πλήρω, αλλά δεν μπορεί και να αποκλειστεί. Όμω η ΕΦΣΑ διατείνεται και η ΕΚΑ, που είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών, θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία όσον αφορά το συσχετισμό με την καρκινογένεση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η εξολόγηση για τους κινδύνους για την υγεία έχει πάρα πολλά προβλήματα και κενά. Αυτά που είδαμε είναι ότι η αξιολόγηση κινδύνου για την υγεία που ετοιμάστηκε καταρχάς από τη γερμανική υπηρεσία BFR βασίζεται κατά πολύ σε εκθέσεις που έχει χρηματοδοτήσει η βιομηχανία. Και ίσως και η Μονσάντο να έχει συγγράψει ε, κάποια από αυτά τα κείμενα. Όσον αφορά αδημοσίευτες μελέτες της βιομηχανίας που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η IARC, ε, είδαμε ότι οι πυρογνώμες Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν έχουν αξιολογήσει όλα τα στοιχεία που είναι παρόντα στις μελέτες της βιομηχανίας, αλλά βασίστηκαν εκτενώς επί της ερμηνείας της βιομηχανίας επί των στοιχείων. Σαν αποτέλεσμα αυτού, σημαντικά πορίσματα έμειναν εκτός της αξιολόγησης ΕΚΑ και της ΕΦΣΑ και οι οργανισμοί το έχουν παραδεχθεί αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις δημοσιευθήσεις ε, μελέτες, είδαμε ότι οι προγνώμε της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αντέγραψαν ουσιαστικά την αξιολόγηση της βιομηχανίας στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεν υπάρχει κάποιο σημάδι ανεξάρτητης αξιολόγησης των μελετών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, εκ, μέρου των πολιτών που είναι πάνω από ένα εκατομμύριο, ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει απαγόρευση όσον αφορά τη γλυφωσάτη κατανοούμε ότι δεν είναι μόνη τη που θα πάρει την απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η πρωτοβουλία των πολιτών εργαλείο που απευθύνεται προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί και θα έπρεπε να προτείνει απαγόρευση της γλυφωσάτη βάσει των περιβαλλοντικών κινδύνων που έχουν αποδειχθεί και που η ΕΦΣΑ και η ΕΚΑ έχουν αναγνωρίσει βάσει της επιστημονικής αβεβαιότητας όσον αφορά τις συνέπειες για την υγεία, κυρίως το συσχετισμό με, την, με τον καρκίνο, εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και θα έπρεπε να εφαρμόσει την αρχή της ε, πρόληψης. Και τρίτον, και άλλοι παράγοντες θεμητοί μπορούν, μπορούν να ληφθούν υπόψη και ζητούμε, και δεν εντάσσεται επίσημα στην πρωτοβουλία μας αυτό, διότι όταν συντάσαμε την πρωτοβουλία δεν περιμέναμε πάνω τόσο άσχημα τα πράγματα, όμως ζητάμε τους λαμβάνοντας την απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσουν τα ρυθμιστικά κενά που διαπιστώθηκαν από την αξιολόγηση κινδύνου. Ευχαριστώ. Στα μέλη του Κοινοβουλίου τώρα θα δώσουμε η κυρία Αγιούσο. Ε, δύο λεπτά ο καθένας. Ναι, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που οργανώνετε αυτή τη συνάντηση. Ακούστε, εδώ μας παρουσιάσατε, ε, μαζεύετε υπογραφές στο κέντρο των πόλεων. Εγώ αν πάω στο κέντρο οποιαδήποτε πόλη και πω ότι η ασπιρίνη σκοτώνει, θα αρχίσουν να υπογράφουν. Έχετε συλλέξει ποτέ όμως ε, ε, υπογραφές στη, στην Ήπεθρο με τους γεωργούς. Ξέρετε ότι η γλυφοσάτη οδηγεί στο να έχουμε λιγότερη καταστροφή της γης. Ε, να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση της ενέργειας, ε, της ε, καλλιέργειας, να μην χρησιμοποιείται υπερβολική, ε, να μην χρειάζεται μεγάλος κόπος και ανθρώπινο δυναμικό για, τα, για να μπορέσουμε να εκτιζώσουμε τα, τα, τα ζωνιοκτώνια. Ακούστε, υπήρξαν πολλέ εκθέσει. Μα πρόσθεσε μια έκθεση. Πολλές όμως επιστημονικές άλλες άλλε εκθέσει. Είχαμε η ΕΦΣΑ, από τι ΗΠΑ, αρμόδια Επιτροπή, η αρμόδια Επιτροπή για την Αξιολόγηση Κινδύνου, το Υπουργείο Γεωργίας ε, της, ε, των ΗΠΑ, η FDA στις ΗΠΑ. Κανείς δεν είπε ότι είναι καρκινογόνο. Κανείς. Μας είπαν ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα για τα ζώα και όχι για τους ανθρώπους. Και στη συνέχεια ε, αποδείχθηκε ότι όλες αυτές οι εκθέσεις ήταν απολύτως διαφανής. Η μόνη που δεν ήταν διαφανής, η μόνη έκθεση ήταν η ERC. Μάλιστα υπάρχουν, το IRC, υπάρχουν μάλιστα τρεις επιστήμονες, η IRC, ο κύριος Τζέιμσον και ο κύριος Μπλερ, που είπαν ότι στις, στα πρώτα σχέδια έκθεσης αναφερόταν κάποια επιστημονικά στοιχεία που λέγανε ότι η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνα. Και στη συνέχεια αυτό αποσύρθηκε από την τελική έκθεση. Δεν μπορείτε να μας τα εξηγήσετε όλα αυτά. Γιατί πολλοί κόσμοι ξέρουν τη γλυφοσάτη. Να σας πω κάτι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας με τη Μονσάντο. Αν δεν την είχε βάλει στην αγορά τη, τη, τη Μονσάντο δεν θα, ήμασταν εδώ ε, σήμερα για να ζητούμε να αποσυρθεί. Και δεν είμαι, έχω καμία, καμία φιλική προτιάση προς τη Μονσάντο. Ευχαριστώ η κυρία Ντάλι, τώρα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους ε, της πρωτοβουλίας πολιτών. Είναι ενδιαφέρον, διότι στο Κοινοβούλιο υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Εγώ εκπροσωπώ τη σοσιαλιστική ομάδα, σοσιαλιστές και δημοκράτες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και όπως είπατε, και εσείς γνωρίζετε τις τελευταίες, το τελευταίο ψήφισμα του Κοινοβουλίου τον περσμένο μήνα όπου δεν συμφωνήσαμε με την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανανέωση της γλυφοσάρης για τα επόμενα 10 χρόνια. Ζητήσαμε σταδιακή ε, ε, απόσυρση έως το 2022 και ζητούμε βεβαίως ε, άμεση χρήση για μη ε, επαγγελματικούς χρήστες. Άμεση απαγόρευση, συγγνώμη. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίω ότι πρέπει να δώσουμε μια μεταβατική περίοδο, να δώσουμε χρόνο στους επαγγελματίε, στους γεωργού στον κλάδο για να προσαρμοστεί. Όμως συμφωνούμε με κάποιε από τις ανησυχίε που εκφράσατε. Η έλλειψη διαφάνειας, το θέμα της, ε, του κατά πόσο τα στοιχεία είναι αξιόπιστα και το θέμα της επιστημονικής ανεξαρτησίας. Στην παρουσίαση σας και εσείς υπογραμμίσατε ε, ότι υπάρχει ένα θέμα ε, σχετικά με την αξιολόγηση, διότι βασίζεται σε μελέτες που προκύπτουν σε περιοδικά και σε επιστημονικά περιοδικά που ε, η ίδια, ο ίδιος ο κλάδος, η ίδια βιομηχανία ε, χρηματοδοτεί. Είναι πραγματικά λόγος ανησυχίας αυτός, όχι μόνο για τους πολίτες, αλλά και για τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ε, θα ήθελα να επικεντρωθώ αυτό που λέτε εσείς. Εσείς ζητείτε απαγόρευση της Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται ότι ο κλάδος θα το αντικαταστήσει με κάποια άλλη ουσία, με άλλα τοξικά συστατικά. Τι θέλετε όμως να πετύχετε τελικά, διότι απαγορεύοντας την γλυφοσάτη τώρα και εφόσον δεν έχουμε την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης, αυτό επηρεάζει και το δεύτερο μέρος, ε, θα έχουμε άλλες τοξικές ουσίες που θα εμφανιστούν. Ποιο είναι λοιπόν ο στόχο σα, μακροπρόθεσμα ε, σε ό,τι αφορά τι ουσίε αυτέ. Και ένα δεύτερο ερώτημα στα γρήγορα, πώς σκοπεύετε να ρυθμίσετε την παραγωγή και την χρήση ε, της, ε, του προϊόντος αυτού, αφού υπάρχουν ακόμα χώρες που μπορούν να εισάγουν αυτό το προϊόν. Μάλιστα, κυρία Γκέρλινγκ το έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θερμό καλωσόρισμα στα μέλη της Επιτροπής. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, γνωρίζετε ότι η μελέτη της IARC που αναφέρατε τόσο συχνά αντιβαίνει στο βάρος των επιστημονικών στοιχείων. Η ΕΦΣΑ, η ΕΚΑ είναι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εκτός αυτού η κοινή συνεδρίαση για την Ανεθεώση των παρασιτοκτόνων και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Μηχανισμός Υγείας ανήκουν σε αυτούς που δεν συμφωνούν με την IARC ότι η γλυφοσάτη είναι καρκινογόνος ουσία. Δεν συμφωνούν. Γιατί λοιπόν επιμένετε για αυτή τη γενική ε, προσέγγιση ότι είναι καρκινογόνος ουσία. Δεύτερον, αναφέρθηκε ότι οι πολίτες ανησυχούν, διότι αν τους κάνετε έλεγχο ούρων θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει γλυφοσάτη στα ούρα τους. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που στηρίζει αυτό τον ισχυρισμό. Δεν αναφέρεται ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τις μετρήσεις είναι τόσο ακριβείς αυτή την εποχή που θα βρείτε πάρα πολλά στα ούρα σας. Και δεν είναι αναλογική αυτή η δήλωση χωρίς ε, παράθεση στοιχείων. Είναι κάτι ανεύθυνο. Δεύτερον ή τρίτον, δοθησών των προσπαθειών, των φοβερών που έχουν καταβληθεί για την ε, πρωτοβουλία. Από τη WeMove.org βλέπουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει από τη σελίδα. Περίπου ένα εκατομμύριο λοιπόν μέλη υπάρχουν και αυτοί κινητοποιούν την όλη προσέγγιση για να φτάσετε το 1,3 εκατομμύρια ενώ δεν θέλω να υποβαθμίσω τα 1,3 εκατομμύρια ανθρώπων που ανησυχούν και πολύ γιατί να μην ανησυχούν άλλωστε λόγω της παραπληροφόρησης δεν θεωρείτε ότι, Ευρω... ότι... θεωρείτε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε λένε ότι πρέπει να απαγορευτεί η γλυφοσάτη. 1,3 εκατομμύρια είναι λιγότερο από 0,3% του πληθυσμού του γενικού τη Ευρώπη Και με λυπή επιστημονικά στοιχεία θέλετε να απαγορεύσουν η γλυφοσάτη. Γιατί, εξηγήστε το ότι είναι λογικό. Είναι λογικό, είναι υπεύθυνο. Thank you. Uh, ε, Mr. παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Νομίζω ότι είναι πάντοτε καλό να βλέπουμε τι πιστεύουν οι ψηφοφόροι μας. Επίσης αυτό τονίζει ότι φυσικά όλοι θέλουν να μειώσουν τις ποσότητες χημικών, συνθετικών ή οργανικών στη γεωργία. Ό,τι και να είναι το χημικό θα πρέπει να είναι η τελευταία λύση και να χρησιμοποιείται βιώσιμα. Έτσι λοιπόν έρχομαι και στο ερώτημά μου. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων είναι η εξής. Η κατάργηση αυτών των χημικών είναι πραγματικά η απάντηση για το μετασχηματισμό του συστήματός μας και για την ε, ε, να μην υπάρχουν πλέον χημικά. Ε, δεν, ξέρω ότι, ε, δεν ξέρω αν αυτό θα είναι η λύση. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε το σύστημά μας, να εξαρτώμαστε λιγότερο, να έχουμε καλύτερες εναλλακτικέ που ενέχουν λιγότερους κινδύνους. Αυτό λοιπόν το θέμα δεν είναι απλό. Είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις που έχουν γίνει μία. Πρώτον, είναι, υπάρχει πιθανότητα καρκινογένεσης. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Ε, έχουμε ένα σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει κάτι τέτοιο. Αν είναι κάτι καρκινογόνο πρέπει να το απαγορεύσουμε, αν όχι. Δεν υπάρχει επιχείρημα να μην διοδοτηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δεύτερη συζήτηση έχει να κάνει με τη βιώσιμη χρήση αυτών των χημικών. Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως σε αυτό το θέμα και όχι απλώς να απαγορεύσουμε ένα χημικό, το συγκεκριμένο χημικό λέγοντας ότι είναι καρκινογόνο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν έχουμε τη σωστή συζήτηση ξεκινήσει για αυτό το θέμα και σας ρωτάω εσάς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόρφμαμαν, ε, καταρχάς να σας ε, συγχαρώ που ξεκινήσατε αυτή την πρωτοβουλία πολιτών. Εγώ έχω ασχοληθεί πολλές φορές ε, με τέτοιες πρωτοβουλίες και ξέρω πόσο δύσκολο είναι κανείς ε, και να ε, συζητήσει το θέμα αλλά και να συλλέξει όλες αυτές ε, τις ε, υπογραφές, να ξέρει ένα σωστός αριθμός. Το 2009 ξεκίνησε αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά πρέπει να τον χρησιμοποιούμε. Τώρα, επί της ουσίας, νομίζω ότι η αδειοδότηση των ε, χημικών θα πρέπει να γίνεται βάσει επιστημονικών κριτηρίων και όχι λόγω κάποιων ε, δημόσιων εκστρατιών. Θεωρώ λοιπόν ότι η αδειοδότηση των ε, φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη είναι λίγο επιφανειακή μέσω της ΕΦΣΑ. Βλέπετε πόσα παρασιτοκτόνα έχουν αδειοθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τελικά αποσύρονται Βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και στην ιατρική, για να υπάρχει καλύτερη επιχειρηματική δράση, ε, χρησιμοποιούνται κάποια τέτοιες, κάποιες τέτοιες ουσίες. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εάν αυτή η μελέτη είναι ε, όχι μόνο αντικειμενική, αλλά έχει αντιμετωπίσει και κάποιες ε, δυσκολίες. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε ακούσει στην γερμανική τηλεόραση φρικτές ιστορίες ε, για παιδιά που δεν γεννήθηκαν λόγω κάποιων χαπιών ε, ήταν πρόορες ας πούμε εκτρώσεις ε, και υπήρχε και η γλυφοσάτη μέσα σε, αυτό, σε αυτή τη συζήτηση. Μετά μπήκε και στη συζήτηση για τον ιό Τσίκα. Η γλυφοσάτη είναι ένα ζυζανιοκτόνο και δεν πρέπει να φτάσει στο ε, φυτό. Όταν φτάσει στη μιλιά ή σε οποιοδήποτε άλλο τέτοιο δέντρο π.χ. στην ουσία ε, πρέπει να σταματήσει εκεί, δεν πρέπει να μπει στην αλυσίδα διατροφής. Αλλιώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Έτσι λοιπόν έρχομαι στο ερώτημα δεν θεωρείτε ότι το Κοινοβούλιο έχει ξεκάθαρη ευθύνη για το πώς ε, θα γίνονται οι προτάσεις και για το κατά πόσο θα πρέπει ε, να απαγορευτεί αυτή η ουσία. Είναι δική μας ευθύνη για το αν θα φύγουμε από τη γλυφοσάτη στα επόμενα δέκα χρόνια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ε, συγχαρώ αυτή την πρωτοβουλία πολιτών διότι δείχνει ότι όπως το κύριο κ. είναι ζωντανή η δημοκρατία μα. Ναι, υπάρχει, είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, υπάρχει αντιπαράθεση και το αποτέλεσμα τη πρωτοβουλία αυτή ε, μα το δείχνει. 1,3 εκατομμύρια ε, πολίτες, έτσι, είναι πολύ, πολύ ανεύθυνοι. Ε, ο καθένα λοιπόν από εμά πρέπει να σεβαστεί την θέση του καθένα των Ευρωπαίων πολιτών που εξεφράστηκε. Και βεβαίω υπάρχει αντιπαράθεση, διότι ε, μετά τα Monsanto Papers και μετά την αντιπαράθεση στι ΗΠΑ δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε δεν μπορούμε να αναρωτιόμαστε όταν ε, ήδη κάποιοι έχουν θεωρήσει ότι είναι κακινογόνο προϊόν ε, όπως στην Καλιφόρνια. Ε, δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε εμείς ως πολιτικοί θύνοντες. Θέλω να επανέλθω στην περίπτωση της Αργεντινής που ακόμα αυτή τη Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκύριακο ε, είχαμε αποκαλύψεις ότι στις μεγάλες πορές όταν ε, ε, έχουμε, αυτό οδηγεί σε πολλέ ε, ε, ασθένειες οι οποίε δεν έχει ακόμα ξεκριβωθεί ε, πόσο σοβαρέ είναι και πόσο οφείλονται στη λιφοσάτη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ρόλο τη Ευρώπη πρέπει να είναι να δείξει το παράδειγμα. Πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή τη προφύλαξη. Δεν μπορούμε να ανανεώσουμε αυτό το προϊόν. Αυτό άλλωστε αποφασίσαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προστατεύσουμε του 500 εκατομμύρια συμπολίτε μα. Απέναντι ε, ε, στο γεγονό ότι οι πολίτε ε, της Ευρώπη, ε, έχουν όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι μια ευκαιρία για μας να δείξουμε ότι η Ευρώπη ασχολείται με τους συμπολίτε της και του προστατεύει από την υπερπαγκοσμιοποίηση και, τα, και τις πολυεθνικές. Θα πρέπει να επενδύσουμε, διότι υπάρχουν λύσει αγρονομικέ απλές για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας συνοδεύσει προς την κατεύθυνση αυτή και να μας πει ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα ε, σαφώς ε, να, πώς θα βγούμε από την κλειφωσάτη. Όχι άμεσα, αλλά τα επόμενα χρόνια να, ε, να βγούμε από αυτό, να, να, να καταργήσουμε αυτό το προϊόν και να βρούμε άλλες λύσεις. θα πρέπει λοιπόν από κοινού να γίνει μια έρευνα για να δώσουμε τα κατάλληλα στοιχεία τα οποία θα είναι αληθή και αδιαφυσβήτητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κονέτσινα τώρα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία αυτή. Ε, αυτό είναι μόνο ένα μέρος του παζλ. Βέβαια, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχουμε κάνει πολλά σχόλια, έχουμε εκφράσει πολλές φορές τις αντιρρήσεις μας και το βασικό ζήτημα είναι ότι δεν μας ακούει κανείς, δεν μας ακούτε. Ε, εννέα κράτη-μέλη ε, θέλουν να ε, πάυσει η χρήση της ούτε, ούτε αυτά τα εννέα κράτη-μέλη ακούστηκαν ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι μόνο οι πολίτες, είναι και τα κράτη-μέλη τα ίδια που το ζητάνε. Θα πρέπει λοιπόν να ακούσουμε τους συμπολίτε μας, θα πρέπει να τους προστατεύσουμε, είναι δική μας ευθύνη είναι καθήκον μας. Δεν συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι η γλυφοσάτη ε, δεν αποτελεί μέρος ε, των, της διατροφής μας. Ε, το είπε κάποιος από τη Γερμανία. Στην πύρα που πίνετε, στη Γερμανία υπάρχει γλυφοσάτη. Εφόσον λοιπόν υπάρχει η παραμικρή υποψία ότι αυτές οι ουσίες είναι βλαβερές, πρέπει να δράσουμε. Τι κάνουμε όμως εμείς, τα αγνοούμε τα δεδομένα, τα γεγονότα και ψάχνουμε επιχειρήματα για να μην δράσουμε, για να μην αναλάβουμε δράση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ε, επιχειρήματα για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να κάνουμε τα πράγματα αλλού, όχι να μην κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν επαρκείς μέθοδοι αγρονομικές για να ακολουθήσουμε μια διαφορετική οδό, για να προλάβουμε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε ε, τι πολυεθνικέ εταιρείε που θα χρησιμοποιήσουν ε, τέτοιε ουσίε και ακόμα χειρότερε. Υπάρχουν νέε μέθοδοι, ναι, που χρησιμοποιούνται σε πολλά κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε χωρί να χρησιμοποιήσουμε ενδεκτόνα στη γεωργία μα. Θα πρέπει οι πολίτε, οι γεωργοί να ενθαρρυνθούν να ακολουθήσουν αυτή την οδό. Σα ευχαριστώ για την πρωτοβουλία αυτή. Πάντω ε, είναι μία από τι πολλέ ε, που ανοίγουν, μα ανοίγουν τα μάτια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Φόντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε 1,3 εκατομμύρια υπογραφέ και έχουμε δικονοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το 80% των πολιτών είναι κατά τη χρήσης τη. Συμφωνούμε. Πρέπει, όσο πιο γρήγορα απολευθερωθούμε από αυτήν και τόσο καλύτερα. Πρέπει να είμαστε και ρεαλιστέ, να δούμε πραγματικότητα. Σε 25 μέρε εκπνέει η περίοδο αδειοδότηση. Έχουμε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που ζητά την πλήρη απαγόρευση με σταδιακή εξάλληψη σε μια πενταετία και έχουμε τα κράτη-μέλη που δεν έχουν μια οριστική θέση ε, στους διάφορους φορείς. Προς τη μία κατεύθυνση στην άλλη. Λοιπόν, θα πρέπει να το ελέγξουμε αυτό, να κλείσουμε ίσως το τελευταίο κεφάλαιο της γλυφωσάτης στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να έχουμε το φόβο να χάσουν οι γεωργοί τα πάντα. Διότι λέμε ότι όπω θέλει τα, τα πολλά χάνει και τα λίγα, λέμε στην Ιταλία. Θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλύτερο θα ήταν όμω να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία για να έχουμε απόλυτη βεβαιότητα ότι η γλυφωσάτη χρησιμοποιείται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση από μια στιγμή και μετά. Τις τελευταίες εβδομάδες κάποιες πολιτικές δυνάμεις επίσης εθελοντικά δημιούργησαν σύγχυση περιγράφοντα το phasing out σαν μια ανανέωση, κάτι που τεχνικός και διανοητικός είναι ασφαλμένο ε, και διάφορε ΜΚΟ επέκριναν το μέτρο. Λοιπόν, η σταδιακή εξάλληψη οδηγεί στην πλήρη απαγόρευση και δεν θα δοθούν άλλε ανανεώσει και παράτασε. Πραγματική και σύντομη ανανέωση θα άνοιγε όμω διαφορετική προσέγγιση όπου η γλυφοσάτη θα μπορούσε να αδειοδοτείται επανειλημμένα. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που σήμερα θα πρέπει να αποφύγουμε με πάση δυνάμει είναι ανανέωση έστω και ετησίω και να βασιστούμε ε, στην, ε, στο άνοιγμα της διεξόδου. Να έχουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για το τέλος χρήσεως της λιφοσάτης που θα είναι μια νίκη και όχι ήττα. Είναι ιστορική στιγμή και πολυεθνικές όμως ε, προσπαθούν να βρουν δικαιολογία να παρουσιαστούν ως μάρτυρες δεν μπορεί να αρνηθεί αυτή την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ολομέλεια το εγκρίναμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην υποκρίνεται ότι γίνεται τίποτα, να αγνοήσει υπογραφέ όλων αυτών των Ευρωπαίων πολιτών, να αγνοήσει και την άποψη του Ευρωκοινοβουλίου και να αγνοήσει και τα κράτη-μέλη που τελικά βρίσκουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αλλά δεν καταλήγουν σε κάποια οριστική θέση. Ο κύριο Πόρτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μέλη της Επιτροπής των Πολιτών. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, ευχαριστώ για την πρωτοβουλία και ευχαριστώ και όλους εκείνους που υπέγραψαν την πρωτοβουλία που είναι σημαντική. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη. Αναφέρθηκε ότι το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα επ' αυτού του θέματος. Η Μάρια Μντάλη, η εξότιμη συνάδελφος, επανέλαβε αυτά που ζητούμε εμείς Απλούστατη ερώτηση. Θα δεχόσασταν εσείς σαν εκπρόσωπος της Σαν εκπρόσωπο πρωτοβουλία των πολιτών δεχόσαστε το, την, ε, το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που υποστηρίχθηκε από το, τους περισσότερους ε, από τις περισσότερες ομάδες του Κοινοβουλίου για τα καρκινογόνα. Αναφερθήκατε στις καρκινογόνες συνέπειες της ουσίας. Υπάρχουν αμφιβολίες, υπόνοιες κλπ. για τα, τη σχέση αιτίου και αιτιατού σαν φάτον τον καρκίνο. Λάβατε υπόψη και άλλα στοιχεία και άλλες συνέπειες ε, της γλυφοσάτης που ε, χρησιμοποιείται και σαν αντιβιωτικό. Δεν συζητήθηκε καθόλου αυτό. Επίσης ε, εμποδίζει το σχηματισμό και περίπλοκων πρωτεϊνών που βρίσκεται και στα ανθρώπινα κύτταρα. Λάβατε υπόψη και άλλες παρενέργειες της γλυφοσάτης εκτός από την καρκινογένεση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο Σπεντιτσίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα είναι η μέρα σημαντική. Οι εκπρόσωποι των πολιτών στο Κοινοβούλιο αντιμετωπίζουν τους άλλους εκπροσώπους των πολιτών εκείνους που πρότειναν αυτή την πρωτοβουλία που όλοι επικροτούν σήμερα. Και γι' αυτό απευθύνομαι στους συναδέλφους ευρωβουλευτές. Έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις των θεσμικών οργάνων που αναφέρθηκαν, των οργανισμών, το ΙΑΡΚ. E και εκεί αναφέρεται ότι είναι καρκινογόνος το γλυφωσάτι και έχουμε την ΕΦΣΑ και την ΕΚΑ για αυτούς τους φορείς πιθανότατα, όχι σίγουρα, πιθανότατα δεν είναι καρκινογόνος ουσία. Άρα ποτέ δεν συζητήθηκε το θέμα της καρκινογένεσης. Υπάρχει προφανή έλλειψη στοιχείων επιστημονικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα αυτά πρόταση, ε, έκανε πρόταση ανανέωση τη αδειοδότηση για άλλα 10 χρόνια. Και ήταν αντίθετο το Κοινοβούλιο. Όλοι γνωρίζαν ότι η αξία τη αντίρρησή μα θα ήταν απλώ συμβολική. Πολιτική αξία είχε. Και όμω οι βουλευτέ μπλοκαρίστηκαν. Κόλλησαν σε μια διαπραγμάτευση για να καταλήξουν στον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό. Αυτό ελπίζαν. Ποιο είναι ο καλύτερο συμβιβασμό έναντι μια ουσία που πιθανότατα είναι καρκινογόνο, Επτά χρόνια είναι καλύτερα από δέκα. Πέντε χρόνια είναι καλύτερα από επτά. Οι πολίτε πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ο τόπο εκεί όπου μια ουσία απαγορεύεται μέχρι τώρα, μέχρι ότου αποδεικνύεται ότι δεν είναι καρκινογόνο. Γι' αυτό το λόγο εμεί προτείναμε μια τροπολογία με την πλήρη απαγόρευση και άμεση απαγόρευση χρήση τη γλυφοσάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να πω σε εκείνους που προωθούν την πρωτοβουλία ότι αυτή η τροπολογία μας απερίφθη από τους περισσότερους ευρωβουλευτές. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα ότι στην τρίτη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρεται καθόλου η απαγόρευση τη μέσα σε πέντε χρόνια όπως ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο. Αναφέρεται ανανέωση για άλλα πέντε χρόνια της χρήσεως. Λοιπόν, κάτι είναι σίγουρο. Εδώ κάποιο ε, κράτησε το ανάστημά του όρθιο, ενώ πολλοί βουλευτέ που είναι παρόντε ε, δεν έλαβαν υπόψη την κίνησή σας που εκπροσωπείτε τους ε, πολίτες. Η κυρία Χάζενκαμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρωτοβουλία ε, και τους εκπροσώπους της πρωτοβουλίας για την απαγόρευση της γλυφοσάτης Έχουμε πάρα πολλούς υποστηρικτές, ε, πάνω από 3 εκατομμύρια σε όλα τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε λοιπόν πόσο ευρεία είναι η υποστήριξη, όχι μόνο στις πόλεις, αλλά και στις αγροτικές περιοχές. Ε, θέλουμε λοιπόν ε, η Κομισιόν να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνει επέκταση της αδειοδότησης της γλυφοσάτης μέχρι να αντιμετωπιστεί σωστά η πρωτοβουλία των πολιτών. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Τίμερμανς, δεν μπορεί απλώς ε, να ε, παραβλέψει αυτά που ε, γίνονται ε, και δεν είναι καν εδώ για να ακούσει τι έχουν να πούν οι εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας. Είναι σκανδαλώδες θα έλεγα. Η Κομισιόν θέλει να πιέσει προς την κατεύθυνση της επέκτασης της αδειοδότησης για άλλα πέντε χρόνια αρνούμενη της βλάβ, την βλάβη που γίνεται στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον όπως και στα φυτά και στα ζώα. Η Επιτροπή θέλει τελικά να προστατέψει την βιοπικιλότητα ε, και ε, από την χημική βιομηχανία ή απλώς ε, θέλει να προστατεύσει τη βιομηχανία. Βλέπουμε ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη ζητούν απαγόρευση ή στα γρήγορη σταδιακή κατάργηση της γλυφοσάτης, ε, γιατί φαίνεται ότι περνάει στο περιβάλλον, στην τροφή μας, ε, στον οργανισμό μας. Οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως η γλυφοσάτη δεν είναι μόνο καρκινογόνος, αλλά πολύ πιθανόν να παίζει και ρόλο ε, στην επιδείμνωση της αντιμικροβιακής αντοχής. Έτσι λοιπόν, ε, δεν πιστεύετε κι εσείς ότι θα έπρεπε ήδη από σήμερα να καταργηθεί πλήρως η γλυφοσέτη. Ο κύριος Άνιου. Ελπίζω όταν τίθενται αυτά τα ερωτήματα στους πολίτες να τους θυμίζουν ότι μπορεί να είναι σύμφωνα με τον ΠΟΕ καρκινογόνος ή γλυφοσάτη, αλλά ο Πόη λέει ότι και το να κόβουμε τα μαλλιά μας ε, είναι ε, καρκινογόνο ή να κάθεσαι μπροστά στη φωτιά πολλή ώρα ή να δουλεύεις νυχτερινή βάρδια. Επίσης, ο καφές ε, μπορεί να έχει ακόμα περισσότερο η καρκινογόνο δράση. Επίσης, όταν πίνεις καφέ δεν πίνεις γλυφοσάτη. Αναφέρθηκε η αρχή της πρόληψης. Αυτό μάλλον αν υπήρχε όταν εφευρέθη ο ηλεκτρισμός, δεν θα είχαμε καν ηλεκτρισμό. Νομίζω ότι αυτό το υλικό υφίσταται εδώ και 40 χρόνια, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, όλο αυτό το διάστημα οι πολίτες εκτίθεντο σε αυτή την ουσία και δεν υπήρξε ε, κάποιο πρόβλημα. Αυτοί που χρησιμοποιούν ε, το προϊόν ε, συμπυκνωμένο έχουν χίλιες φορές μεγαλύτερη έκθεση. Άνθρωποι όπως η γεωργή, η φυτοπαραγωγή και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ούτε και απόδειξη ότι βλάπτεται η υγεία των ανθρώπων. Αν καταργήσουμε αυτήν την ουσία, οι γεωργοί θα πρέπει να καλλιεργούν όλο και πιο συχνά τη γη. Τέσσερις φορές το χρόνο, για παράδειγμα, για να τάξουν τα ζυζάνια. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της εκπομπής του διοξιδίου του άνθρακα. Ε, οι περισσότεροι από εσά είστε κατά της αύξησης των εκπομπών του διεξιδίου του, του άνθρακα. Ε, επίσης ε, ε, υπάρχει αύξηση διάβρωσης του εδάφους και θα δείτε και όλο περισσότερους γλάρους να έρχονται πίσω από αυτούς που οργώνουν, να τρώνε τους σπόρους και στην ουσία το πρόβλημα θα είναι πλέον οι γλάροι. Επίσης, έχουμε εισαγωγές από χώρες του κόσμου που δεν έχει καταργηθεί η γλυφοσάτη. Πώς θα γίνει ε, λοιπόν. Ε, νομίζω ότι η όλη η ιστορία αυτή είναι μίσος προς μια συγκεκριμένη εταιρεία τη μοσάντο ε, το οποίο σοβεί εδώ και 20 χρόνια. Τέλος η κυρία Όκαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Επιτροπή Αναφορών εδώ. να πω πέρα από την ε, πρωτοβουλία ότι υπάρχουν και νέα αναφορές ε, στην Επιτροπή μας για τη Γλυφοσάτη. Ας ε, σας δείξω μια άλλη οπτική γωνία λοιπόν που έχει να κάνει με την Επιτροπή Αναφορών. Είναι η έλλειψη διαφάνειας και σύγκρουση συμφερόντων. Όταν κάνατε την προσωμείωση μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών ε, οργανώσεων πραγματικά με εξεπλήσαξατε. Ε, αν βλέπατε τι ακριβώς ε, έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος κατά της Μονσάντο, θα καταλαβαίνατε πόσα χρήματα παίζονται. Δεν θα δίσταζα να μιλήσω και για δωροδοκία. Νομίζω λοιπόν ότι το να επιτιθέμεθα στον ΠΟΗ ε, έτσι δεν είναι Σωστό. Όταν έχουμε λοιπόν αμφιβολίες για την πλήρη διαφάνεια, ε, πρέπει κάτι να κάνουμε. Το να έχουμε πλήρη διαφάνεια δεν σημαίνει να κάθεται κάποιος σε μια ε, φωταγωγημένη αίθουσα, ε, ακόμα και η σύγκρουση συμφερόντων είναι τεράστιο ε, πρόβλημα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον ΕΦΣΑ. Γιατί πραγματικά υπάρχουν χρήματα που καταβάλλονται και είναι και μεγάλη η ζημιά που θα αντιμετωπίσουν οι γεωργοί αν υπάρξει απαγόρευση. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την αρχή της ε, πρόληψης η οποία υπάρχει στη συνθήκη αλλά θα πρέπει ακόμα περισσότερο οι πολίτες και το κοινοβούλιο να μπορούν να ε, ε, έχουν μια συζήτηση βάσει μιας διαφανούς διαδικασίας. Όλοι να μπορούν να ε, συνεισφέρουν σε αυτή τη συζήτηση και επιστήμονες που δεν έχουν σχέση με τα χρήματα αυτά ε, για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από ό,τι έχουμε τώρα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα και πάλι το λόγο στην κυρία Άχτερμπεργκ για 15 λεπτά για να απαντήσει στα ερωτήματα των μελών. Ευχαριστούμε για τα ενθαρρυντικά σχόλια από κάποιους ευρωβουλευτές, αλλά και για τις επικρίσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά. Έχουν υποθεί πολλά και έχω 14 ε, λεπτά, 15, 15 λεπτά. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσω με τον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Άγνιου, που μας ε, υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες κατηγοριοποιήσεις ε, ε, καρκινογόνων προϊόντων, το καφές και άλλα προϊόντα. Πρέπει να γίνει εδώ μια, ένας διαχωρισμός. Και άλλοι ευρωβουλευτές είπαν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τον οποίο υπάρχει έκθεση στην γλυφοσάρη. Δεν τον πίνουμε, αλλά εκτιθέμεθα μέσω των τροφίμων, μέσω των ποτών, το νερό. Στο 45% των τη γη τη Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται. Είναι δύσκολο να το αποφύγει, να αποφύγει κανεί την γλυφωσάτη. Ε, έχει εντοπιστεί σε πολλά ε, μέρη, ακόμα και αν δεν το πίνουμε, είμαστε εκτεθειμένοι. Είπατε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ε, καρκίνου για τους γεωργούς. Συγγνώμη, να σας διορθώσω. Η IARC, και θα σας πω μετά για την εμπιστευόμαστε την IARC, λέει ότι υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για τους ανθρώπους μετά από έρευνας, μελέτες, που αφορούσαν γεωργούς. Θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας ε, αυτές οι εκθέσεις. Ε, παρ' όλα αυτά η ΕΦΣΑ, η Μονσάτο ε, θεώρησαν ότι δεν είναι αξιόπιστες. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα περιορισμένα στοιχεία που υπάρχουν για τις, τις βλάβες στην ανθρώπινη υγεία υπάρχουν όμως με βάση αυτή τη μελέτη της IARC Θα ξεκινήσω από την πρώτη ομιλητή, είναι πιο εύκολο νομίζω. Εσείς, ε, κυρία Αγιούσο, αμφισβητείτε ότι οι γεωργοί υποστηρίζουν την απαγόρευση γλυφωσάτης, διότι ε, η γλυφωσάτη έχει πολλά ωφέλη για τους γεωργούς. Να σας θυμίσω ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές οργανώσεις γεωργών. Κάποιες οργανώσεις γεωργών θέλουν να κρατήσουν την γλυφοσάτη. Δεν θέλουν να την εγκαταλείψουν, παρότι είναι στην πρώτη γραμμή και παρότι υπάρχουν κάποια λίγα στοιχεία καρκίνου στους γεωργούς λόγω της γλυφοσάτης, χρήσης γλυφοσάτης. Υπάρχουν όμως και οργανώσεις ε, γεωργών που κατάλαβαν, έχουν αντιληφθεί ότι αυτή η, ουσία πρέπει να αποσυρθεί και είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης αυτής. Όχι μόνο έχω καταλάβει ότι πρέπει να καταργηθεί, σκέφτονται ήδη ποιες θα είναι οι λύσεις ε, για τους γεωργούς, χωρίς την γλυφοσάτη. Αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει και χαιρόμαστε που αυτό συμβαίνει και μεταξύ των γεωργών δύο οργανώσεις, έτσι, μία στη Γαλλία και μία στη Γερμανία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Ισπανία. Επίσης, οι ευρωβουλευτές μας θύμισαν και τις άλλες αξιολογήσεις που έγιναν ανά τον κόσμο, όχι μόνο από την ΕΦΣΑ και την ΕΚΑ, που είπαν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ε, για την, ε, τον καρκινογόνο χαρακτήρα της λιφοσάτης να σας θυμίσω γιατί εμείς επισκεφτήκαμε την IARC. Η IARC είναι μια εξαιρετικά σεβαστή υπηρεσία με πολύ αυστηρούς κανόνες, πολύ αυστηρά πρότυπα. Εργάζεται με διαλεγμένους εμπειρογνώμονες, γνωστούς με το όνομά τους και που δεν έχουν εξαρτήσεις. Και επίσης εργάζεται μόνο με δημοσιευμένα δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα έχει μεγάλη φήμη. Το Μάρτιο του 2016 περίπου 100 επιστήμονες έγραψαν ένα κείμενο που υπερασπίζεται τις 100, την, κατηγοριοποίηση ε, της ε, IARC και λέγοντας ότι οι εκθέσεις της ΕΦΣΑ παρουσιάζουν πολλά, προγράμματα, πολλά προβλήματα. Επίσης γίνεται περάσπιση του συνολικού προγράμματος της IARC. Ε, να, να υπενθυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη επίθεση που δέχεται η IARC από τη χημική βιομηχανία. Υπάρχει μια άλλη εκστρατεία από την ε, βιομηχανία καπνού. Μετά την κατηγοριοποίηση ε, περικαρκίνου σε ό,τι αφορά ε, τους καπνιστές. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν ικανοποιούνται ε, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα υψηλά, τα υψηλά πρότυπα, τι υψηλέ προδιαγραφέ, να αποφύγουμε τη σύγκρουση συμφερόντων τα άτομα τα οποία έχουν εξαρτήσει. Αυτό υποτίθεται ότι προβλέπει ήδη ο μηχανισμός ο συμβουλευτικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εργάζεται μόνο με δημοσιευμένα στοιχεία. Βεβαίω ο κλάδο, δεν, δεν, δεν θα, η βιομηχανία δεν θα είναι ικανοποιημένη, αλλά για να μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη και να υπάρξει αξιοπιστία και μεταξύ τη επιστημονική κοινότητα και με του πολίτε, αυτό είναι ο δρόμο. Επίση, δύο μιλητέ μα κατηγόρησαν ότι όλα αυτά αφορούν τη Μονσάντο. Δεν έχει σχέση με την κλειφωσάτη. Είναι επειδή αυτή η συγκεκριμένη πολυεθνική ε, είναι αυτή η οποία έβαλε στην αγορά την, την γλυφοσάτη. Γνωρίζουμε ότι η γλυφοσάτη παράγεται από 20 διαφορετικές εταιρείες και όχι μόνο η Μοντσάντο. Πολλοί πιέζουν για την αντιδότηση της γλυφοσάτης. Βέβαια η Μονσάντο παίζει έναν ηγετικό ρόλο σε αυτήν την ε, ομάδα λομπιστών που ζητούν ανανέωση της άδειας. Είναι στην πρώτη γραμμή αυτοί είναι που κάνουν προσπάθειες στον επιστημονικό κλάδο, στη δημόσια συζήτηση. Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τη Μοντσάτο όταν μιλάμε για τη γλυφοσάτη, εν περιπτώσει. Τι θέλουμε να πετύχουμε, ρώτησε η κυρία Ντάλη. Η απαγόρευση της γλυφοσάτης ε, ενδεχομένως να, να έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν άλλες τοξικές ουσίες που θα την και τι ε, θα έχουμε πετύχει αν τελικά εισάγουμε τη γλυφοσάτη όχι ως προϊόν αλλά ως κατάλοιπα ε, στα εισαγόμενα, ε, στις εισαγόμενες οτροφές. Βεβαίως και δεν θέλουμε η γλυφοσάτη να κατασταθεί από κάτι άλλο από κάποιο άλλο τοξικό ζανιοκτόνο. Επίσης, δεν θεωρούμε ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Και είμαστε κάπως αισιόδοξοι, να σου πω και γιατί. Δεν θα συνεχίσει η ίδια απειλή χωρίς τη γλυφωσάτη. Η γλυφοσάτη είναι ένα ζενιοκτόνο ε, το οποίο είναι συνολικό, είναι ολικό. Ε, είναι, δεν υπάρχει αντικατάσταση για αυτό το προϊόν τώρα. Ξέρουμε ότι χρησιμοποιείται και από δημόσιες αρχές, από εταιρείε, από τους ιδιώτες. Αδείγματος χάρη, το γλυφόσανάιτ, που είναι ο ανταγωνιστής, ας πούμε, της γλυφοσάτης, το, το λέει και ο Επίτροπος Ανταγωνισμού της Ένωσης, δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη μαζικά, έχει περιοριστεί λόγω των επιπτώσεων για την υγεία. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα παρόμοιο, με παρόμοια χημική ουσία έχει επιβεβαιωθεί από προβολές, προβλέψεις ε, των γεωργών ε, που αποδεικνύουν στο μέλλον θα χρησιμοποιούν λιγότερα ζανιοκτώνα και θα πληρώνουν λιγότερα χρήματα για ζανιοκτώνα οι γεωργοί. Γι' αυτό ανησυχεί και ο κλάδος. Γι' αυτό και επιμένει τόσο πολύ και γαντζώνεται από την κλειφωσάτη. Η εναλλακτική τώρα. Και αυτό το δείχνουν οι προβλέψεις. Είναι να αλλάξουν οι γεωργικές πρακτικές. Και αυτό είναι ακόμα κάτι το οποίο δεν θέλουν οι χημικές, η χημική βιομηχανία, διότι θα χάσουν χρήματα. Ένα άλλο λόγο για τον οποίο είμαστε αισιόδοξοι, ότι δεν θα είναι δηλαδή η ίδια η, ίδια η ζημιά ε, χωρί τη γλυφωσάτη, είναι ότι ε, τα έχουμε ξανακούσει αυτά τα επιχειρήματα. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μερικώ απαγόλησε τρία νε, νεονικοτινοειδή, είχε πει, ε, είχαν, έλεγε τότε ο κλάδο ότι θα έρθουν άλλα χημικά που θα την καταστήσουν και θα συνεχίσουν οι βλαβερέ συνέπειε και ότι δεν θα υπάρξει βελτίωση. Σήμερα όμω, το 2016 έχουμε στοιχεία από τον Εμένο Βασίλειο που δείχνουν ότι η χρήση των εντομοκτώνων ε, δεν αυξήθηκε μετά την απαγόρευση των νοικοτινοειδών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, ότι δεν ήρθαν να αντικατασταθούν τα νεονικοτινοειδή από, άλλες, από άλλα προϊόντα, άλλα ζανιοκτώνα. Δεν αυξάνεται η κατανάλωσή τους, η ζήτησή τους. Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άλλα βλαβερά ζανιοκτώνα και καλό είναι να μην τα χρησιμοποιούν οι γεωργοί. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που υπάρχουν τρία αιτήματα τρει στόχοι. Θα αναφερθεί και η Αγγελική συνάδελφο την Τρίτη, που είναι η συνολική μείωση τη χρήση των ζενιοκτώνων και των εντομοκτώνων, των παρασιτοκτώνων στην Ευρώπη. Για να έρθω τώρα στη Judy Girling, Julie Gerling και τα σχολιά τη. Το γεγονός ότι η γλυφωσάτη έχει βρεθεί στα ούρα είναι προβληματικό. Γιατί? βεβαίω μιλάμε για μικρές, μικρή περιεκτικότητα, μικρή ποσότητα, αλλά υπάρχει στο σώμα μας αυτό, ε, αυτή η ουσία και αν είναι τοξική τότε δεν υπάρχει κάποιο επίπεδο ασφαλείας, δεν υπάρχει κάποιο κατόφλι κάτω από το οποίο είμαστε ασφαλείς. Δεν είναι πάντα ζήτημα ποσότητας. λέτε ότι 0,3% του πληθυσμού μας υποστηρίζει, ακούστε, έχουν γίνει μελέτες, ο Μίκα αναφέρθηκε προηγουμένως, έχουν γίνει δημοσκοπήσεις 70, 80, 78% του πληθυσμού ε, ε, σε πέντε κράτη-μέλη της Ένωσης υποστηρίζουν ε, την απαγόρευση της γλυφοσάτης, οπότε είμαστε πολύ, μιλάμε για μεγέθη πολύ μεγαλύτερα από αυτών που υπέγραψαν τις υπογραφές. Αυτό ήταν το όριο, το 1 εκατομμύριο, μαζέψαμε 1,3 εκατομμύρια και μετά ήρθαμε και φέραμε την πρωτοβουλία εδώ. Δεν, δεν συνεχίσαμε γιατί δεν υπήρχε λόγος. Να έρθω τώρα σε αυτό που είπε ο κύριο ε, Χάιτιμερ. Η απαγόρευση των χημικών είναι απάντηση. Λύνει τα προβλήματά μας. Βεβαίως και δεν τα λύνει. Είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι να δώσουμε μια ρυθμιστική απάντηση, μια επίπεδο ρυθμίσεων απέναντι στον κίνδυνο. Το αποτέλεσμα και το το πιστεύουμε αυτό και για την απαγόρευση της γλυφοσάτης, αλλά και για άλλες απαγορεύσεις χημικών. Θα πρέπει να είναι αλλαγή στις γεωργικές πρακτικές. Είναι κάτι που συμβαίνει ήδη. Ο Μίκα αναφέρθηκε σχετικά. Χιλιάδες ε, βιολογικές καλλιέργειες ε, δουλεύουν χωρίς γλυφοσάτη και μη, γεωργικές, και μη βιολογικές καλλιέργειες. Αυτές οι βελτιώσεις ε, στις γεωργικές πρακτικές, πρακτικές θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν ο κανόνας, έτσι ώστε όλοι οι γεωργοί να μπορούν να την ακολουθήσουν. Βεβαίω αυτό προποθέτει περισσότερη δουλειά, περισσότερε γνώσει, περισσότερη πραγματομοσύνη για του γεωργού. Κάποιοι ειδικοί είπαν ότι αυτή η διαθεσιμότητα ε, αυτού του φτηνού ζανιοκτώνου έχει ε, παρεμποδίσει την καινοτομία. Η καινοτομία ε, και οι εφευρέσεις προκύπτουν από την ανάγκη. Όσο θα υπάρχει σαν το δεν θα έχουμε καινοτομία. Είναι φτηνό, είναι διαθέσιμο, θα το χρησιμοποιούν οι γεωργοί. Όταν λοιπόν αυτή η ουσία απαγορευτεί, να αναμένεται και περισσότερες θέσεις απασχόλησης στη Γεωργία και περισσότερη καινοτομία στη Γεωργία. Και ένα σημαντικό στοιχείο θα πρέπει να, μια, να συνοδεύσουμε, να βοηθήσουμε τους Γεωργούς για να συμβούν αυτά τα πράγματα. Εσείς εδώ, οι ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτήν την ε, κατηγορία ότι η καμπάνια αυτή είναι επιφανειακή και ότι χρησιμοποιούμε δεδομένα τα οποία δεν είναι ε, επιβεβαιωμένα. Το είπε ο κ. Ντόρφμαν αυτό. Εμείς είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, αναφερθήκαμε ε, σε στοιχεία, σε ευρήματα επιστημονικά, χρησιμοποιήσαμε την έκθεση της IARC, γιατί είναι αξιόπιστη η IARC, εξηγήσαμε, εξήγησα γιατί εμπιστευόμαστε την IARC και δεν νομίζω να υπήρξε καμία, ε, κανένα επιχείρημα αστήρικτο σε ό,τι αφορά τη Και ναι κύριε Ντόρφμαν, πιστεύουμε ότι είναι και υπεύθυνο και είναι ένα πολύ καλό βήμα η, η απαγόρευση της χρήσης ε, της γλυφοσάτης πρώτης σποράς. Διότι μένουν, μένουν κατάλοιπα στα φρούτα. Έγινε αναφορά προηγουμένω σε πρόσφατες ε, έρευνες. Ναι, πρέπει να συνοψίσετε σιγά σιγά. Αναφέρθηκε σε νέα ευρήματα που δείχνει ότι η γλυφοσάτη, η έκθεση στη γλυφοσάτη μπορεί να υπονομεύσει τη χρήση αντιβιωτικών και την, ε, της, ε, τη δράση των αντιβιωτικών. Αυτή είναι άλλη μια μελέτη που έχετε να δείξει πώς ανησυχητικά είναι τα πράγματα όχι μόνο με τη γλυφοσάτη βέβαια, αυτό ισχύει και για άλλα ζανιοκτώνα. Η μελέτη όμως αυτή λέει κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ακολουθήσουν μια ευρύτερη προσέγγιση. Το τι είναι ασφαλές και τι είναι σωστό να χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη έχει αλλάξει με το καιρό και πρέπει να αλλάξει και άλλο. Να αλλάξει ξανά για να λάβουμε υπόψη μας τέτοιου είδους ανησυχίες διότι η αντιμικροβιακή αντίσταση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και για σας κύριε Επίτροπε πρέπει να αποτελέσει και αυτό μέρος της αξιολόγησης ε, κινδύνου για τον ζανιοκτώνων. Κλείνοντας, να πω ότι όλα αυτά τα σχόλια ήταν εξαιρετικά χρήσιμα και σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη ο κ. Πότς μας θύμισε ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε απαγόρευση γλυφοσάτης, ε, μια μερική απαγόρευση τώρα και πλήρη απαγόρευση σε 5-10 χρόνια. Χαιρόμαστε για αυτή τη θέση του Κοινοβουλίου. Η δική μας θέση και η θέση που εκπροσωπεί εδώ και η Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ότι η γλυφοσάτη πρέπει να απαγορευτεί τώρα. Θεωρούμε ότι η θέση του Κοινοβουλίου είναι προϊόν πολιτικού συμβασμού και είναι και η πιο προοδευτική θέση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ε, και ελπίζουμε αυτό να οδηγήσει σε ένα τελικό συμβασμό στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σαμπίνα Γιούλικερ αρμόδια για την ασφάλεια τροφίμων και φυτών και καινοτομία τη Γενική Διευθύνσεω για την Υγεία DG Santa. Ένα πεντάλεπτο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω αφετηρία τη ανταλλαγή απόψεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι και η αξιολόγηση κινδύνου και η έγκριση της γλυφοσάτης υπόκεινται σε διαδικασίες και κριτήρια που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί παρασιτοκτόνων που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και, το Ευρωκοινοβούλιο. Οι διατάξεις της νομοθεσίας συμπεριλαμβάνουν την προστασία της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Να τονίσω ότι οι διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας εδράζονται επί της αρχής της προλήψεως. Η αρχή της πρόληψης είναι ένα απόσπαστο τμήμα των διατάξεων της εν λόγω νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι μετά την υποβολή και αξιολόγηση αίτηση για ανανέωση ενεργού συστατικού, όπως είναι η γλυφοσάτη, η νομοθεσία υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει δεόντως. Να εθετήσει δηλαδή τον κανονισμό είτε μέσω ανανεώσεως της εγκρίσεως ενεργού ουσίας υπό όρους ή να μην ανανεώσει την έγκριση της εν λόγω ουσίας. Πιο συγκεκριμένα, η νομοθεσία τι προβλέπει ανανέωση της εγκρίσεως ενεργούσιας εάν τα κριτήρια εγκρίσεως πληρούνται. Στη ρυθμιστική διαδικασία όσον αφορά την γλυφοσάτη δεν είδαμε να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Βέβαια υπάρχει εδώ και το ερώτημα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγορεύει τη γλυφοσάτη και δεν προτείνει κάτι τέτοιο. Υπήρξαμε σαφείς. Δεν υπάρχουν λόγοι επιστημονικοί ή νομικοί για την απαγόρευση της γλυφοσάτης στα πλαίσια της νομοθεσίας για τα παρασιτοκτόνα που προανέφερα. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που υπευλήθη και εκπρόσωποι αυτής αναφέρθηκαν σοβαρές απειλές για την ανθρώπινη υγεία ισχυρίζονται ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Η γλυφοσάτη ανεξαρτήτως και διεξοδικά αξιολογήθηκε από τα κράτη-μέλη, από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τις Χημικές Ουσίες. Και το συμπέρασμα ήταν το ίδιο σε κάθε περίπτωση. Ταξινόμηση της γλυφοσάτης που δεν δικαιολογείται να ταξινομηθεί γλυφοσάτη ως καρκινογόνος ουσία και η αξιολόγηση κινδύνου τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπέρανε ότι η γλυφοσάτη, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τι ορθέ γεωργικέ πρακτικέ, δεν δημιουργεί απαράδεκτου κινδύνου για του ανθρώπου, για τα ζώα, ούτε για το περιβάλλον. Και οι εθνικέ αρχέ άλλων νομοθεσιών, όπω είναι ο Καναδά, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, και η συνεδρίαση του ΦΑΟ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία για τα Παρασυτοκτόνα και είναι αυτή η συνεδρίαση κατά συμπεράματα. Η IARC, ο Διεθνή Φορέα για την Έρευνα για τον Καρκίνο, είναι ο μόνο οργανισμό που έχει αποκλίνουσα άποψη όσον αφορά ε, καρκίνογόνε συνέπειε τη γλυφοσάτη. Βλέποντα λοιπόν τον έλεγχο των πληροφοριών για τη γλυφοσάτη, αναλύοντα προσεκτικά τι διαθέσιμε πληροφορίε. και μετά διεξοδική ανάλυση. Επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος αμφισβητήσεως της επιστημονικής εξολογήσεως και των σχετικών πορισμάτων γλυφοσάτη που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω του συστήματος που δημιούργησε για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, ενεστώτος έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στα κάτι μέλη πρόταση για ανανέωση τη εγκρίσεως της εν λόγω για μια πενταετία. Να πω κάτι άλλο Κάτι που ακούστηκε θέλω να αναφέρω όσον αφορά τη σταδιακή εξάλληψη της γλυφοσάτης. Να σας πω ότι η ισχύουσα νομοθεσία και οι προναφερθέντες όροι δεν προβλέπουν οριστική ημερομηνία για την ε, πάυση χρήσεως της ουσίας, για την απαγόρηση της ουσίας. Όμως, μια ανανέωση της δραστικής αυτής ουσίας επιτρέπει κάτι άλλο και ζητεί μάλλον κάτι άλλο. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη εντό ενός έτους πρέπει να επαναξιολογήσουν την αδειοδότηση όλων των προϊόντων στην αγορά τους. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους συμπληρωματικούς όρους που καθορίστηκαν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παραδείγματος χάρη. Προστασία υπογείων υδάτων, η χρήση της ουσίας σε δημοσίους χώρους πρέπει να γίνεται προσεκτικά, όπως και η χρήση πριν από το θερισμό και συλλογή του καρπού, πριν τη συγκομιδή. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της ανανέωσης της αδειοδοτήσεως για την ουσία. Τελειώνει ο χρόνος μου. Αυτό που είπε η κυρία Άουκεν. Από ό,τι κατάλαβα, αυτά που είπε η κυρία Άουκεν, νομίζω ότι κάτι είπε όσον αφορά την ευρωπαϊκή αξιολόγηση που υπόκειται σε δωροδοκία από ό,τι κατανόησα. Απορρίπτω αυτό τον ισχυρισμό εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη υποφαινομένη και των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Άχτεμπεργκ αν έχετε κάποια σύντομα σχόλια σχετικά με αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μονολεκτικά, μάλλον σε μία φράση. Δεν έχετε πολύ χρόνο. Σε μία φράση θέλω να πω ότι είναι άδικο η απόφαση για τη γλυφοσάτη και, τα προϊόντα που περιέχουν γλυφοσάτη να αφήνεται στα κάτι μέλη. Γιατί, διότι η ΕΦΣΑ είπε ότι αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα από την ίδια την γλυφοσάτη. Αυτό κατέδειξαν και ανεξάρτητε μελέτε που πραγματοποιήθηκαν. Η ΕΦΣΑ λέει ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση. Το θέμα είναι τα κράτη-μέλη πώ θα αξιολογήσουν αυτό το κίνδυνο. Έχουν στοιχεία. Δεν υπάρχουν απαιτήσει για στοιχεία για προϊόντα ξεχωριστά για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι καρκινογενή, έχουν καρκινοτοξικότητα κλπ. και μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία. Δεν αξιολογούνται αυτά τα προϊόντα. Μονσάν το είπε ότι δεν το κάνει. Είναι μια εταιρεία που αποφάσισε να απορρίψει αυτές τις ανησυχίες των πελατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να απορρίψει τις ανησυχίες. Αυτός είναι ένας όλος λόγος να απαγορευτεί η γλυφωσάτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο των συζητήσεων. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στο δεύτερο στόχο της πρωτοβουλίας, αλλαγές δηλαδή στην επιστημονική αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα παρασιτοκτόνα. Για την παρουσίαση των λόγων στόχου έχουμε τον κύριο Helmut Bulcher, εκπρόσωπο της Επιτροπής των Πολιτών Χωρίς να χρονοτριβήσουμε λοιπόν, σας δίνουμε το λόγο για ένα πεντάλεπτο. Καλημέρα. Καταρχάς να σας χαιρετήσω όλους. Ε, ονομάζομαι Χέλμουτ ε, Μπούρτσαρ, είμαι βιοχημικός ε, και εργάζομαι για το Friends of the Earth. Είμαι υπεύθυνο ε, για την γλυφοσάτη, για τις διαδικασίες αδειοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το, ε, για τα λάθη, τα ξεκάθαρα λάθη του συστήματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη το 2009 έδωσαν άδεια για ένα νέο, ε, έβγαλαν ε, μια οδηγία για τα ζυζανιοκτώνα που μιλάει για την ειδική προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας. Ε, αυτή η προσέγγιση προβλέπει ε, οι καρκινογόνες ε, ε, ουσίες, μεταλλαξιογόνες, ουσίες λοιπά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ε, παρασιτοκτόνα. Και αυτό πάντοτε λαμβάνοντα υπόψη την επιστημονική βιβλιογραφία. Οι δημοσιευμένες μελέτες, ε, οι οποίες δηλαδή προέρχονται από αντικειμενικούς ε, επιστήμονες δείχνουν ότι η ανανέωση της άδειας της γλυφοσάτης, η οποία ήδη από το 2013 φαίνεται σε αντίστοιχη έκθεση ότι προφανώς να έχει καρκινογόνο δράση, ε, αν ε, παραμείνει λοιπόν η αδειοδότηση θα υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτό είμαστε τώρα εδώ διότι η γλυφοσάτη αποτελεί ε, παράδειγμα ε, ενός ε, σοβαρού σφάλματος του συστήματος αδειοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματα που οι υπεύθυνοι έχουν αγνοήσει, έχουν διαψεύσει και τελικά δεν ελήφθη υπόψη η επιστημονική βιβλιογραφία. Για να δούμε, ας πούμε, μια μελέτη η οποία μιλά για τις βλαπτικές επιπτώσεις της γλυφοσάτης. Η επιστημονική βιβλιογραφία μιλάει συγκεκριμένα για αυτές τις βλαπτικές επιπτώσεις της γλυφοστάτης σε τρεις-τέσσερες ε, ε, μελέτες. Ε, το κέντρο για τη μελέτη κατά του καρκίνου του ΠΟΗ είχε βγάλει το ίδιο συμπέρασμα. Επίσης, η πρώτη αξιολόγηση ε, ή όταν έγινε η πρώτη αξιολόγηση υπήρχαν ήδη μελέτες ε, από τους παραγωγούς και εκεί φαινόταν ε, ότι τα, τα στοιχεία δεν ήταν σχετικά ούτε πιστικά. Το BFR, το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Αξιολόγηση των Κινδύνων, ε, δεν έκανε αντικειμενική αξιολόγηση αυτής της μέλωτης σύμφωνα με το άρθρο 11 της αντίστοιχη οδηγίας ε, όπου λέει ότι πρέπει να έχουμε και τις αξιολογήσει των επιστημόνων και τις διάφορες ερμηνείες ε, στην έκθεση για την αξιολόγηση ενός προϊόντος. Δεν υπήρξε καν σχόλιο για αυτά. Υπάρχει μια έκθεση 46 σελίδων, την έχω εδώ μαζί μου, η οποία δείχνει ότι στην ουσία ε, σε τέτοιες ε, πολύ σημαντικές περιπτώσεις έγινε μόνο ένα copy-paste και υπάρχουν ε, διάφορα κίνητρα να μεταφερθεί η ευθύνη σε μέρη τα οποία έχουν σύγκρουση συμφερόντων. Τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν δώσει την εντολή για να γίνουν μελέτες που περιγράφουν τα προϊόντα τους ως μη βλαπτικά. Έτσι λοιπόν, ε, πέρα από αυτό, ε, να πούμε ότι οι μελέτες αυτές ε, δεν δίνονται και στον δημόσιο, στη δημόσια συζήτηση λόγω των εμπορικών, της εμπειρικής εμπιστευτικότητας. Υπάρχουν ε, λύσεις όμως για αυτά τα προβλήματα, οι οποίες ε, στην ουσία είναι τρεις τροποποιήσεις ε, που ζητά και η πρωτοβουλία. Πρώτον, να σταματήσει η σύγκρουση συμφερόντων που, υπάρχουν, που υπάρχει λόγω των εργαστηρίων οποία, στα οποία ανατίθεται συγκεκριμένα η μελέτη αυτή. Θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές οι οποίες στην ουσία θα ελέγχουν ε, την επιστημονική ποιότητα ε, των στοιχείων. Δεύτερον, κάθε ε, ρυθμιστική μελέτη θα πρέπει να δημοσιοποιείται. Θα πρέπει να υπάρχει ένα έξτρακτ, ε, μια σύνοψη στις διάφορες βάσεις δεδομένων και μέσα από αυτή να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στα raw data. Ε, έτσι λοιπόν οι μελέτες αυτές θα μπορούν να είναι κομμάτι της επιστημονικής συζήτησης. Και τρίτον, οι αρχές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και δεν θα πρέπει να γίνεται στρατηγική επιλογή των αρχών στις οποίες απευθυνόμαστε στο μέλλον. Όταν γίνουν αυτά τα βήματα νομίζω ότι το ευρωπαϊκό σύστημα αδειοδότησης θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ευρώπης. Και αυτό θα είναι μια καλή αρχή νομίζω. Ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο στους βουλευτές ε, η κυρία Γκίζεκε είναι η πρώτη που θέλει να πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Ο κύριος Γκίζεκε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο κύριος Στούτσικ έχει κάνει ε, μία ανακοίνωση ε, σε μία γερμανική εφημερίδα που λέει ότι... Ε, ο, κύριος ε, ε, αυτός έχει πάρει 1.600 δολάρια ε, από κάποιους επιστήμονες. Το, η, αυτή, αυτό το κέντρο για τον καρκίνο συγκεκριμένα έχει πληρώσει χρήματα. Άρα ε, αυτούς τους επιστήμονες πρέπει να τους λάβουμε σοβαρά υπόψη μας αν παίρνουν λεφτά από δικηγορικά γραφεία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αντικειμενική να απαντηθεί παρακαλώ αυτό το ερώτημα. Και δεύτερον, ως προς τη διαδικασία, έχει να κάνει και με τη γλυφοσάτη και ε, με όλα τα στοιχεία στα οποία χρειάζονται επιστημονικά στοιχεία. Η δόση πάντοτε ε, δημιουργεί το δηλητήριο, λέγεται, λέμε συνήθως. Άρα πρέπει να υπάρξει μια αντίστοιχη μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη και το μέγεθος του κινδύνου. Ε, η δυναμικότητα του κινδύνου είναι πολύ σημαντική. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε ε, συναισθηματικές συζητήσεις εδώ. Πρέπει να, να, να κοιτάμε αντικειμενικά την επιστήμη και να κάνουμε αντίστοιχα τις εκτιμήσεις μας. Ευχαριστώ κυρία Κάντενμπαχ. Ευχαριστώ πολύ και ακούστε για την απάντησή σας και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Πραγματικά ήταν ε, εξαιρετικά εντυπωσιακό σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να μαζεύσετε τόσες ε, υπογραφές, 1,3 εκατομμύρια και δεν ήταν ότι απλά μιλούσατε στις, στα κέντρα πόλη και μαζεύετε υπογραφέ, και είναι κάτι πολύ περισσότερο. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τη συμμόρφωση με τις ε, διαδικασίες που, που είναι εγκεκριμένε. Ιδιαίτερα το 8.5 του κανονισμού, έτσι ώστε ε, να υπάρχει εξολόγηση ομοτήμων και να ανησυχεί αυτό. Συμφωνείτε ότι η επιστημονική εξολόγηση ομοτήμων πρέπει μόνο αυτή να λάβει υπόψη, να υπόψη στην λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, συμφωνείτε ότι ο κλάδος θα πρέπει να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία στην ΕΦΣΑ και αν υπάρχουν σημαντικά κενά η ενεργή ουσία να μην εγκρίνεται. Πριν τελειώσει ο χρόνος μου θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μέρος του Ευρωκοινοβουλίου διότι είμαι βέβαιη ότι είμαστε το πιο διαφανές κοινοβούλιο στον κόσμο. Δεν είμαστε βεβαίως ομοιογενείς ε, στις θέσεις μας, ε, όπως διαπιστώσατε και σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να δείτε ποιος ψηφίζει τι σε αυτό το κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα όταν αποφασίζετε για τις επόμενες ευρωεκλογέ του Ευρωκοινοβουλίου το 2019. Πραγματικά κοιτάξτε τι έκαναν εδώ οι βουλευτές στο Κοινοβούλιο, ποιος ψήφισε τι. Διότι είμαστε εδώ για να εκπροσωπήσουμε τα δικά σας συμφέροντα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ε, το Κοινοβούλιο, είναι ο κάθε βουλευτής που εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρώπης. Ψηφίστε λοιπόν για τα μέλη, για τα μελλοντικά μέλη που θα εκπροσωπούν τα, τα δικά σας συμφέροντα ε, και τη δική σας ε, γνώμη. Ναι, ελπίζω όντως να συμβαίνει αυτό το ποιος ψηφίζει τι, πραγματικά το ελπίζω. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, η κυρία Γκροστέτ έχει το λόγο τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ αντιλαμβάνομαι βεβαίω ότι υπάρχουν επιφυλάξεις, υπάρχουν κριτικέ επικρίσεις ε, σε ό,τι αφορά το σύστημα αδειοδότηση ε, τις μελέτες ε, που υποβάλλονται με τα προβλήματα σύγκρουση συμφερόντων. Το αντιλαμβάνομαι απολύτω. Πρέπει όμω να πούμε και στη θέση των βουλευτών. Όταν ακούμε εμπειρογνώμονε, συνήθω μετά ξέρουμε ακόμα λιγότερα διότι πάντα υπάρχει κάποιο εμπειρογνώμο που δεν συμφωνεί με τον άλλον. Ε, είναι περίπλοκο. Πρέπει να βασιστούμε λοιπόν στι ε, υπηρεσίε, στου οργανισμού. Τώρα βέβαια μετά υπάρχει κριτική από του οργανισμού, την ΕΦΣΑ, την ΕΚΑ. Ε, και εδώ πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια δουλειά, να δώσουμε μεγαλύτερα, περισσότερα μέσα σε αυτέ τι υπηρεσίε για να μπορούν να είναι παντελώ ανεξάρτητε. Όταν μιλάμε όμω για συγκρού συμφερόντων, πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Διότι εφόσον ε, απομακρύνουν πυρογνώμονε με το πρόσχημα ότι μπορεί να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ε, χάνουμε την ποιότητα τη πραγματογνωμοσύνη κάποιων εμπειρογνωμόνων. Και να πούμε ότι η πραγματογνωμοσύνη μπορεί να προέρχεται από τον κλάδο, ε, να το απαγορεύσουμε αυτό. Ε, και αυτό λάθος είναι, διότι ο κλάδος γνωρίζει τα προϊόντα, έχει πραγματογνωμοσύνη και μπορεί να μιλήσει για αυτά εμπεριστατωμένα. Θα ήθελα λοιπόν να επιστρέψω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ναι, βεβαίως, ίσως να πρέπει να ζητήσουμε να ε, μεταρρυθμιστούν, μεταρρυθμιστούν αυτές οι υπηρεσίες για να είναι όσο γίνεται πιο ανεξάρτητες στο έργο τους. Αλλά προσοχή, προσοχή ε, δεν πρέπει ε, να σκεφτόμαστε ιδεολογικά εδώ ε, σε ό,τι αφορά το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόμπες, Λόμπες Μπερμέχο έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε που οργανώσατε αυτή την ε, συνάντηση, την ακρόαση και την αλλαγή απόψεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΦΣΑ βασίζονται σε δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί και δεδομένα που δεν έχουν δημοσιευθεί για την αξιολόγησή του. Η ΕΦΣΑ είπε ότι εξέτασε μελέτες, επιπλέον μελέτες του κλάδου. Μελέτες που δεν έχουν δημοσιευθεί. Για να καθορίσουν ε, ότι για να φτάσουν στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ απίθανο να υπάρξει καρκίνος να εμφανιστεί καρκίνο. Αυτέ οι εκθέσει δεν είναι διαθέσιμε. Παρότι τι ζητήσαμε. Ζητήσαμε να έχουν πρόσβαση, για να τι δούμε, να τι μελετήσουμε. Και όμω πολλέ από αυτέ εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμε. Εξακολουθούν να μην μπορούμε να τι δούμε. Ούτε καν από την IARC. Λοιπόν, τα ερωτήματά μου αφορούν κυρίω στην Κομισιόν. Θα ήθελα να ξέρω έω πότε θα συνεχιστεί αυτή η έλλειψη διαφάνειας για να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις. Θα ήθελα επίσης να ξέρω εάν κάποια στιγμή θα ε, σεβαστείτε την αποφάση του δικαστηρίου που λέει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποκρύπτονται με βάση την, το επιχείρημα του εμπορικού απόρριτου. Ούτε αυτό το σέβεστε. Η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών είναι πάνω από τα συμφέροντα του κλάδου του βιομηχανικού. Έχουμε δει πολλές φορές στο το Κοινοβούλιο πώς, ο κλάδο, πώς η βιομηχανία επηρεάζει τις αποφάσεις που παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως με την πρόσφατη περίπτωση του Dieselgate. Και θα ήθελα να ξέρω επίσης έως πότε θα συνεχίσετε να επιτρέπετε η βιομηχανία να αποφασίζει ποιο κράτος μέλος θα κάνει τις επιστημονικές αξιολογήσεις. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να αλλάξουν. Και κάτι άλλο και τελειώνω. Υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν υπογραμμίσει τις επιπτώσεις της γλυφοσάτης ως ε, ε, ενδοκρινική διατράκτης. Ε, εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε τη δική της νομοθεσία για να, για να καθορίσει επιστημονικά κριτήρια για τις ορμονικούς κινδύνους αυτών των ουσιών. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα λοιπόν, ποιες είναι οι επιπτώσεις της γλυφοσάτης ε, ως προϊόν ενδοκρινικός, ε, διαχείριση. Ε, ακούστε, η ύπεθρος πεθαίνει αυτή τη στιγμή. Εάν θέλετε να βελτιώσετε την παραγωγή, αν θέλετε να υπάρξει καλύτερη χρήση της γης, αν θέλετε να βελτιώσετε την ίδια τη γη, σταματήστε να, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το ζυνοκτώνα και επενδύστε σε, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζούλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για πολλωστή φορά Απευθύνομαι προς τον Επίτροπο τον κύριο Αντρουκάητη. Έχω απλούστατη ερώτηση. Πόσο σημαντική είναι η προστασία της υγείας των πολιτών. Έγινε συζήτηση σήμερα και διεξάγεται μια σημαντική συζήτηση σήμερα. Όπως βλέπω τα πράγματα, ε, μιλάμε για την γραφειοκρατία, περιοριζόμαστε από τα εμπόδια και δεν μπαίνουμε στην ουσία όμως, που είναι η υγεία του περιβάλλοντος και των πολιτών. Μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάτι άλλο σημαντικότατο. Δεν μπορεί να κάνετε κάτι άλλο, λέτε, από να εγκρίνετε την ανανέωση. Καμία στατηγική διεξόδου. Και αυτό που με θλίβει περισσότερο και με κουράζει θα έλεγα και με ενοχλεί είναι ότι μια πλευρά έχουμε κινήματα όπως είναι το δικό μας. Κινήματα των πολιτών που ζητούν την απαγόρευση της ουσίας. Που δεν κάνει καλό. Αυτό είναι γεγονός. Αυτή η ουσία δεν κάνει καλό. Απ' την άλλη, όμως, έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κολλάει στην γραφειοκρατία. Απ' τη μία πλευρά, λοιπόν, έχουμε ένα κίνημα πολιτών, ένα κίνημα των εκλεγμένων θεσμών των πολιτών που εκπροσωπούν τους πολίτες και από την άλλη μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή με άτομα που απαρτίζεται από άτομα που δεν είναι αιρετά και δεν προωθούν τα συμφέροντα των πολιτών. Δεν εκπροσωπούν τους πολίτες. Καταλαβαίνω αυτή την γραφειοκρατική σύγχυση, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Εάν βάλουμε στο επίκεντρο την υγεία, εγώ περιμένω από εκείνον που σήμερα έχει στο χέρι το παιχνίδι να βρει μια πρόταση προς τη προς την έξοδο. Δεν με νοιάζει να μάθω ο, αν δεν υπάρχουν νομικές τεχνικές δυνατότητες που δεν δίνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διακόψει αυτή την πορεία. Θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει στεναρή θέση. Λοιπόν, Επιτροπέ, ρωτώ, αν το Συμβούλιο παραμένει σε αποτελμάτωση και δεν βοηθάει, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα εξακολουθεί να προστατεύεται από την γραφειοκρατία, να, δημιουργεί, ε, να προβάλλει σαν πρόσχημα την γραφειοκρατία. Κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε ήδη διάφορους συναδέλφους. Παρουσίασαν πολλά επιχειρήματα για τη μία ανανέωση διοδότησης της ε, ουσίας. Να διακοπεί αμέσω η διοδότησή της. Να δώσουν απάντηση της Task Force για την γλυφοσάτη που απέστειλε, ε, της οποίας ηγείται η Μονσάντο, που έστειλε αμέσως μετά ψηφοφορία του ψηφίσματος πέρσι του Ευρωκοινοβουλίου. Και έστειλε απάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε είχε το θράσος να πει ότι η συζήτηση είναι σε συναισθηματικό επίπεδο και παράλογο και απομακρυνόμαστε από μια επιστημονική προσέγγιση. Πιστεύω ότι αυτό είναι μεγάλο ψεύδος. Δεν μπορούμε να αμφισβητούμε τη συνεισφορά της ίδιας επιστήμης που προσπαθεί να ρίξει φως σε ένα θέμα πολύ αδιαφανές και σκοτεινό. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις τρέχουσες ερεύνες και από τα δικαστήρια των ΗΠΑ και από το σκάνδαλο Monsanto Papers. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Να μην βλέπουμε ότι πλευρά σε επιστημόνων ότι χρησιμοποιούν οι εταιρείε αυτές και επιστήμονες για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Είναι παλιό παρασιτοχτόνο η γλυφοσάτη είχε εγκριθεί τη δεκαετία του 70 και τη χρησιμοποιούμε ακόμα. Έχει προξενήσει φοβερές ζημιές. Εδώ βλέπουμε ένα διάγραμμα και βλέπουμε την εκθετική αύξηση της αντίστασης ε, στα, όσον αφορά τα παράσιτα, τα ζυζάνια, η αντίσταση των ζυζανίων. Δεν είναι σύγχρονη τεχνολογία που σχηρίζεται Task Force της Monsanto. Εδώ μιλάμε για κάτι απερχιωμένο, ξεπερασμένο, που δεν έχει λόγο ύπαρξης. Θα ήθελα ο Επίτροπος να λάβει μια θαραλέα απόφαση, με στένος, και στο τέλος του έτους να απαγορεύσει την χρήση αυτής της ουσίας. Εδώ ολοκληρώσαμε, λέει Πρόεδρος, τις ερωτήσεις των μελών. Ο κ. Χέρμοντ Μπούτσαρ θα δώσει απαντήσεις. 15 λεπτά το πολύ έχει στη διάθεσή του. Ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω με τη σειρά. Η πρώτη ερώτηση από τον κύριο Κίσεγκε είχε να κάνει με την αξιοπιστία της αξιολόγησης του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο, η ΆΡΚ, λέγοντας ότι ο Κρίστοφερ Πορτιέ πήρε χρήματα ε, για να μπορέσει να εκπροσωπήσει ένα αμερικανικό δικηγορικό γραφείο ε, ως ειδικό. Αυτά τα χρήματα τα πήρε εδώ και πάρα πολύ καιρό και γι' αυτό η το ΙΑΡΚ δεν τον είχε συμπεριλάβει στους εμπειρογνώμονες για λόγω αυτής της σύγκρουσης συμφερόντων και συγκεκριμένα στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, ε, με αυτό το θέμα που έσκασε για τη Μονσάντο ε, είδαμε πώς ακριβώς λειτουργεί το αμερικανικό σύστημα με τις ε, μαζικές αυτές ε, μηνύσεις όπου παίρνουμε επιστήμονες οι οποίοι είχαν συμβόλαιο και τους εξετάζουμε για να δούμε για τη σύγκρουση συμφερόντων. Ο Κρίστοφερ Πορτιέ ήταν μεταξύ αυτών. Αυτή λοιπόν η αιτίαση είναι μία από τις πολλές ε, που έχουμε. Και πραγματικά δείχνει ε, ότι δεν μπορούμε να θέτουμε σε αμφισβήτηση την ε, αξιοπιστία του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για το καρκίνο γιατί στην ουσία αντιμετωπίζει εντατικά τέτοιες αιτιάσεις διότι βλέπετε ε, πολλές φορές ε, οι δημοσιογράφοι είναι ασυγκράτητοι, ούτε καν δημοσιογραφία δεν κάνουν. Προσπαθούν λοιπόν να ελέγχουν όλες αυτές ε, τις κατηγορίες. Το IARC λοιπόν έβγαλε από την τελική έκθεση στοιχεία που έλεγαν ότι εδώ δεν βλέπουμε καρκινογένεση. Γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι επιστήμονες που το έγραψαν αυτό ήταν πληρωμένοι από τη Μονσάντο. Ήταν βάση της ε, έκθεσης ε, της έρευνας ε, της Μονσάντο και αν την αφήσουμε αυτή στην άκρη βλέπουμε ότι υπάρχει καρκινογόνος δράση. Επίσης ε, υπήρξε και μια άλλη περιγραφή από μια άλλη μελέτη ε, που είχε πληρώσει η Μονσάντο ε, πάλι από έναν επιστήμονο της δεκαετίας του 80 που δεν είναι αντικειμενικός και αυτός ο οποίος έγραφε αντίστοιχα πράγματα. Αυτά ήθελα να πω στον κύριο Κίσεγκερ. Όμως, ε, με σόκαρε το γεγονός ε, ότι ε, μιλάτε για την οδηγία ε, και λέτε ότι πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το άρθρο σχετικά με την καρκινογένεση. Ε, νομίζω πραγματικά ότι αν οι επιστήμονες θεωρούν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δεν πρέπει να τον αφήσουμε στην άκρη. Γι' αυτό, και το λόγο, γι αυτό το λόγο το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έθεσαν αυτά τα βασικά κριτήρια για τις συγκεκριμένες ιδιότητες. Τώρα η ερώτηση 2 από την κυρία Κάντεμπαχ. η οποία θεωρεί ότι πρέπει ε, να αλλάξουμε τη διαδικασία του peer review της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι αντίστοιχο με τη δεύτερη απέτηση που έχουμε για το σύστημα διοδότησης. Ε, πρέπει να αναγνωρίζονται μόνο μελέτες που έχουν δημοσιοποιηθεί, δημοσιευθεί, αλλά συγκεκριμένα, να είναι έρευνες οι οποίες έχουν συγκεκριμένα δεδομένα και αυτές οι μελέτες να περνάνε το τεστ του κατά πόσο είναι ψευδής ή όχι. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που τις έχει, έχει αναθέσει στα συγκεκριμένα εργαστήρια να κάνουν τις ε, μελέτες. Ε, αν είναι ένα εργαστήριο το οποίο είναι σε ανταγωνισμό με άλλο, ε, και τα λοιπά ε, και να διασφαλίζουμε ότι η μελέτη είναι από ανεξάρτητο εργαστήριο. Το τρίτο θέμα τέθηκε από την κυρία Κατσέτε η οποία ε, είπε συγκεκριμένα ότι πρέπει να βλέπουμε τις απόψεις των επιστημόνων. Ε, είπε ότι επικρίνουμε ε, την ΕΦΣΑ και διάφορες υπηρεσίες ε, και ρώτησε αν αυτό είναι δικαιολογημένο. Ε, κοιτάξτε, πολλές φορές πραγματικά εκπλήσωμε που ποτέ δεν υπάρχει αμφισβήτηση για το κατά πόσο έχουν γίνει σωστές διαδικασίες για κάποιες τέτοιες μελέτες. Όπως είπε και ο κύριος Ανδροκαΐτης, ε, πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη έρευνα. Σύμφωνα με το άρθρο 11, εάν έχει γίνει ανεξάρτητη έρευνα βάσει της επιστημονικής βιβλιογραφίας, ε, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν υπάρχει όμως οποιοδήποτε στοιχείο ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, Ας πούμε στο κεφάλαιο για την ε, γονιδιοτοξικότητα ε, δεν υπάρχει ούτε μία ε, πρόταση που να μην μπορούμε να πηρύψουμε στη Μονσάντο. Πραγματικά έχουν αντιγράψει τα πάντα. Και αν η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο δεν αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, δεν θα κλείσει ποτέ αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει άλλη μία δεύτερη ερώτηση, πολύ ενδιαφέρουσα που έθεσε η κυρία Γκροστέτ, η σύγκρουση συμφερόντων. Ε, συμφωνώ πλήρως μαζί της ότι η σύγκρουση των συμφερόντων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να κλείσουμε αυτή την βιομηχανία. Η βιομηχανία έχει γνώση, αλλά δεν έχει και νόημα να δίνουμε ε, αρμοδιότητες στην βιομηχανία όταν μπορεί αυτές να τις εκτελέσει άνετα μια υπηρεσία ανεξάρτητη. Γιατί ε, είναι αδύνατο να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Φυσικά ως παραγωγός θα πω ότι θα κάνω ανεξάρτητη αξιολόγηση, αλλά θα κλείσω και την εταιρεία μου. Ε, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβούν. Μια άλλη ερώτηση είχε να κάνει με το κατά πόσο η διαφάνεια, το γεγονός ότι οι μελέτες ε, ε, είναι από τους ίδιους τους παραγωγούς των ουσιών ε, ε, έχει νόημα. Αυτό που δεν έχει νόημα είναι να ε, κρατάμε μυστικές αυτές τις μελέτες. Το αναγνωρίζουμε όλοι και εσείς νομίζω και ο Επίτροπος Ανδρουκαίτης το είπε πολύ ξεκάθαρα ότι το ερώτημα είναι κατά πόσο θα πρέπει στο εξής να ανεχόμαστε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η απάντηση είναι καθαρή. Οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες δεν καταλαβαίνουν. Όταν ε, συχνά ταξιδεύω λόγω του βιβλίου που έχω γράψει και ακούω τι λέει ο κόσμος, πραγματικά κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί κρατούν Τιούνται μυστικές αυτές οι μελέτες που εμπεριστατώνουν το ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν μπορεί να συνεχίσει κάτι τέτοιο γιατί η εμπιστοσύνη των πολιτών διαταράσσεται. Και φυσικά υπάρχουν και νομικές συνοεπίες και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Διαδικαστήριο τον Νοέμβριο του 2016 ε, αποφάσισε ότι θα πρέπει όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ζυζανιοκτώνα να είναι δημοσιοποιημένα. Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, να επιμείνουμε σε αυτό. Τέλος, ε, οι δύο τελευταίοι ομιλητές ε, είπαν πράγματα με τα οποία συμφωνώ. Ο κύριος Τσούλα πραγματικά ε, είπε ότι λείπει η συζήτηση επί του περιεχομένου σε αυτό το ζήτημα με την κλειφωσάτη και εμένα μου λείπει αυτή η συζήτηση επί του περιεχομένου με ελάχιστες εξαιρέσεις ε, η συζήτηση δεν περιέχει ποτέ την ουσία. Όταν μιλάμε για την αξιολόγηση κινδύνων, εδώ και δύο χρόνια υφίσταται η φήμη ότι έπρεπε να γίνει μία αξιολόγηση των κινδύνων σύμφωνα, ε, για την καρκινογόνο δράση. Ε, αυτό ε, έπρεπε να το κάνει το, το αντίστοιχο Ομοσπονδιακό Γραφείο για την Αξιολόγηση των Κινδύνων. Υπάρχει αυτή η φήμη τόσο καιρό και δεν την έχει κανείς διαψεύσει. Ε, δεν έχει δοθεί κάποια γραπτή απάντηση. Νομίζω μόνο ότι τον Σεπτέμβριο του 2015 δόθηκε μια απάντηση στην, στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας. Ε, ε, ενώ εξορισμού ε, θα πρέπει η συγκεκριμένη υπηρεσία να χρησιμοποιεί ανεξάρτητες μελέτες και να, και να χρησιμοποιεί τα στοιχεία για την επισήμανση και την ταξινόμηση των χημικών. Εδώ στην Ευρώπη έχουμε αντίστοιχο σύστημα. Μιλάμε για, το, για την ταξινόμηση των κινδύνων σύμφωνα με το, την αξιολόγηση του ΙΑΡΚ. Για να αποφασίσουμε λοιπόν πώς θα ταξινομήσουμε βάσει του κινδύνου ένα χημικό, μια δραστική ουσία, δηλαδή για να δούμε αν είναι καρκινογόνο ή όχι, θα πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία για να πάρει μετά την άδεια. Και αυτό το συγκεκριμένο ε, στοιχείο του κανονισμού 1107 του 2009 είναι που παραβιάζεται εδώ και δύο χρόνια εντατικά. Το ακούω από παντού. Αυτό είναι το θεμελιώδες πρόβλημα. Κανείς δεν μπορεί να ανεχτεί ε, να τα ψεύδη. Τα, τα ψεύδη στην ουσία δεν μας βοηθούν να κάνουμε πολιτική. Και σε μία συνέντευξη του Διευθυντή της ΕΦΣΑ ακούσαμε ότι υπάρχει κίνδυνος για ε, καρκινογένεση. Ε, βέβαια, ε, είπε ότι δεν υφίσταται αυτός στους ανθρώπους. Δεν λειτουργούν έτσι οι νόμοι μας. Να πω τώρα και, να πω και στο τελευταίο σημείο που είναι το ερώτημα πώς ορίζεται η επιστήμη. Γιατί υπάρχει όλο και περισσότερο το επιχείρημα και από τη βιομηχανία και από τις αρχές ότι εδώ έχουμε μία επιστημονική μελέτη και επιστημονικά στοιχεία και πρέπει να αποφασίσουμε. Πρέπει να κοιτάμε τι είδους επιστήμη είναι αυτή όμως. Είναι ένα απλό copy-paste. Είναι κάτι που το έχει ζητήσει η Μονσάντο και βάζει τέτοιε ανοησίες μέσα στην ε, έρευνα ο επιστήμονας. Αν ε, κανείς θέλει να είναι αντικειμενικός θα πρέπει να κοιτάξει στο IARC. Αυτό είναι το Ινστιτούτο το οποίο μπορεί να πιστοποιήσει κάτι τέτοιο γιατί ε, δεν έχει τους επιστήμονες που εκπροσωπούν τη Μονσάντο, γιατί συνέχεια λέμε ότι είναι από τη μία η Μονσάντο και από την άλλη οι επικριτές της γλυφοσάτης που είναι πολύ συναισθηματικοί. Ε, όμως εδώ και πολλά χρόνια έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα και πραγματικά να πω ότι έρχεται η στιγμή να δούμε επιτέλους ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να επεκτείνουμε την αδειοδότηση της γλυφοσάτης βάσει επιστημονικών στοιχείων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπούτσερ και τώρα ε, ο, α, ο κύριος Μίνκο από την Κομισιόν ε, είναι ο αντιπρόεδρος ε, της Γενικής Διεύθυνσης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αντιδράσω τα πέντε λεπτά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν πρόκειται να επαναλάβω ζητήματα που απαντήθηκαν νωρίτερα από τον συνάδελφο στα πλαίσια του πρώτου ερωτήματος. Εδώ Μιλάμε για τη διαδικασία. Για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, με τις μελέτες και πώς ε, αυτές ε, ε, εκπονούνται. Είναι πιο γενικά ζητήματα και βέβαιως εξαιρετικά σημαντικά και για μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα των συμφερόντων. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε ότι ε, εξετάστηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ η παρούσα νομοθεσία. Θεωρήθηκε ε, με νομοθεσία σταθμός. Ε, και αυτή την νομοθεσία ακολουθούμε τώρα. Το βάρος της απόδειξης για την ασφάλεια μιας ενεργού ουσία ή την ουσίας, είτε είναι ζυνοκτόνο είτε όχι, το έχει η εταιρεία. Και ε, αναλαμβάνει και το σχετικό κόστος. Και είμαι βέβαιος ότι αυτός είναι ένα σαφής λόγος ε, για τη συμφωνία που υπήρξε στο Κοινοβούλιο και μεταξύ των συνομοθετών γενικότερα. Πρέπει να πω επίσης ότι είναι το ίδιο σύστημα το οποίο είναι και ευρύτερο, έτσι, αφορά τα φάρμακα, όχι μόνο τα ζενοκτώνα, αφορά πολλά προϊόντα. Τώρα, όταν ζητάει μια έγκριση μια εταιρεία ε, ή μια ανανέωση, πρέπει να υποβάλει τις μελέτες που προβλέπονται στα πλαίσια των διεθνών προδιαγραφών σύμφωνα με τις ορθές εργαστηριακές πρακτικές και τα πρωτόκολλα που προβλέπονται στα πλαίσια των διεθνών προτύπων. Ε, να πω ότι τα θέματα αυτά τα κοιτάζουμε εδώ και καιρό. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα για την εκπόνηση των μελετών τα εργαστήρια ενδεχομένως μπορούν ε, να ε, απομακρυνθούν, να αποκλίνουν για να ικανοποιήσουν αυτό που έχει ζητήσει την έκθεση. Δεν είναι εύκολο αυτό. Ε, τα πρωτόκολλα είναι σαφή. Οι πρακτικές είναι συγκεκριμένες. Είναι δύσκολο να, αποκλίνει κανείς. Βεβαίως από εκεί και πέρα ζητείτε ε, να χρησιμοποιούνται δημοσιευμένα ε, μελέτες, δημοσιευμένη βιβλιογραφία, προϊόν ε, αξιολόγηση ομοτήμων. Αυτό υπάρχει ήδη. Έτσι. Ε, οι μελέτες που υποβάλλει ο κλάδος έρχονται να προσθεθούν σε αυτές που έχουν ζητηθεί ε, νωρίτερα. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα αίτημα σε ό,τι αφορά το πώ θα εκπονούνται και πώ θα ζητούνται αυτές οι εκθέσει. Να πω ότι, και θα ξεκινήσω πρώτα με το θέμα της διαφάνειας και της ενημέρωσης ε, για τα ε, στοιχεία, ε, τα κατέργαστα. Ε, σε αυτή την περίπτωση, εφόσον εφαρμόσουμε την νομοθεσία, ακολουθούμε αυτό που μας ζητάει η νομοθεσία. Δηλαδή, η ΕΦΣΑ να κάνει ε, μια περίληψη που θα είναι δημοσιοποιημένοι, θα υπάρχουν στοιχεία των επιμέρους ε, ε, ερευνών που θα δημοσιοποιούνται και όλα τα ε, έγγραφα τα οποία έρχονται να υποστηρίξουν τη γνώμη της ΕΦΣΑ για την ενεργή ουσία. Όλα αυτά που να δημοσιευθούν από την ΕΦΣΑ. Είναι η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και στην ΕΚΑ. Γνωρίζετε ότι έγινε και μια συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει να δημοσιοποιούνται και τα κατέργαστα δεδομένα. Η ΕΦΣΑ τα μοιράζεται για τους ευρωβουλευτές που το ζητούν, υπάρχει μια αίθουσα κλειστή για την ανάγνωσή τους, όμως βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι εδώ μιλάμε, ζητάτε μια πιο συστημική διαφάνεια, πιο συστημικά μέτρα διαφάνειας. Τα θέματα αυτά δεν είναι καινούρια για μας. Τα συζητάμε εδώ και καιρό. Τα είχαμε ήδη εντοπίσει στις συζητήσεις μας ε, στο, στην REFIT ε, για το γενική νομοθεσία σχετικά με τα τρόφιμα και βεβαίως ε, δεν παραμελούμε, δεν αγνοούμε αυτά, αυτή την έκκληση, προσπαθούμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια και ζητούμε από, από αυτούς που έχουν την πληροφορία στα χέρια τους να, φαν, και αυτοί, να εμπλεκακούν και αυτοί. Τώρα, λέτε πόσο καιρό, για πόσο καιρό θα έχουμε έλλειψη διαφάνειας. Θα εξετάσουμε τις αναλλακτικέ. Ε, νομίζω ότι θα συζητηθούν οι ενδυνάμοι λύσεις όσα αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Να πω κάτι τώρα για τις μελέτες. Διότι νομίζω ότι αυτό το αίτημα να μην βασιζόμαστε στις μελέτες του ετώντα πρέπει να λάβει υπόψη κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιληφθούμε ότι μιλάμε για ένα πολύ μικρό αριθμό μελετών όπου υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Νομίζω ότι πάνω από 95% των μελετών ε, δεν δημιούργησαν καμία αντιπαράθεση. Επιπλέον, ε, να σας πω ότι οι μελέτες που συνδέονται με τις εγκρίσεις ε, στο σύστημα αυτό που εφαρμόζουμε είναι 20.000 μελέτες το χρόνο. 20.000, έτσι. Σας το λέω για να καταλάβετε, να αντιληφθείτε γιατί μεγέθη μιλάμε. Για πόση δουλειά χρειάζεται, για πόση δουλειά χρειάζεται. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οπωσδήποτε. Το κόστος αλλά και η αξιοπιστία βεβαίως. Βεβαίως ε, είναι σαφές με βάση όλα αυτά τα επιχειρήματα ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αντιπρόπωση του προβλήματος. Ψάχνουμε τρόπο βελτίωσης ε, της διαχείρισης ε, της διαδικασίας έγκρισης. υπάρχει ένας έλεγχος διαδικασίας μέσω ελέγχων που θα διενεργούν οι υπηρεσίες, οι οργανισμοί. Ενδεχομένως ε, και η δυνατότητα να ζητηθεί ανεξάρτητη έρευνα. Ιδιαίτερα ε, στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει ε, αντιπαράθεση, διότι σας είπα ότι είναι με λίγες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ και τώρα ο κύριος Μπούρτσερ, δεν ξέρω αν θέλει να αντιδράσει σε αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε ένα λεπτό όμως. Ένα λεπτό, μάλιστα. Zuerst Καταρχάς, χαίρομαι ιδιαίτερα που η Κομισιόν θα ασχοληθεί με το θέμα της διαφάνειας για την αρχή ότι ο παραγωγός πρέπει να αποδείξει ότι είναι ασφαλές ε, το προϊόν του. Η δική μας ε, πρόταση ε, είναι να μην είναι ο παραγωγός ο οποίος θα αναθέτει στο συγκεκριμένο εργαστήριο τη μελέτη, αλλά θα λέει χρειάζομαι μελέτη και θα την αναθέτει σε μια υπηρεσία ανεξάρτητη. Και έτσι δεν θα υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος και η σύγκρουση συμφερόντων. Ο σύνδεσμος με το εργαστήριο δηλαδή. Και τώρα η Κομισιόν δεν ε, ανησυχεί που το 75% της ε, έκθεσης αξιολόγησης μιλά για επιστημονικές μελέτες οι οποίες δείχνουν πως ε, ε, έχει γονιδιοτοξικότητα η γλυφοσάτη 75% όχι 25% και μόνο μία είναι η μελέτη η οποία έχει θετικές αξιολογήσεις έχουμε διάφορους επιστημονικούς κόσμους και μετά οι αρχές εδώ μονομερός ε, ε, ε, ε επαφίονται σε αυτά που έχουν απλώς αντιγραφεί από αυτά που λέει η Μονσάντο. Έτσι είναι. Και είναι πρόβλημα. Και πραγματικά δεν ανησυχείτε. Όποιος δεν ανησυχεί, αν δεν ανησυχείτε πραγματικά δεν καταλαβαίνω πλέον αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστώ. Καλώς ολοκληρώσαμε το δεύτερο γύρο και πάμε στον τελευταίο. Υποχρεωτική μείωση και στόχους για τη χρήση παρασιτοκτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να παρουσιαστεί ο στόχος για την Επιτροπή των Πολιτών. Είναι, είναι η κυρία Αγγελική Λυσιμάχου. Έχετε το λόγο για ένα πεντάλεπτο στη διάθεσή σας. Πέντε λεπτά. Τώρα είναι πέντε λεπτά. Και μετά ένα τέταρτο. Ξεκινάμε με ένα πεντάλεπτο. Για να παρουσιάσετε το στόχο σας. Um, Σας ευχαριστώ. Θα παρουσιάσω τον τρίτο στόχο. Μείωση της χρήσης παρασιτοκτόνων και σχετική στόχος για ένα μέλλον χωρίς παρασιτοκτόνα. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την κλειφωσάτη κοινωνία μας. Εξαρτάται πολύ από τα παρασιτοκτόνα. Και έτσι κάθε χρόνο περίπου 400.000 τόνοι δαστικών ουσιών απελευθερώνονται στο περιβάλλον αυτός ο αριθμός θα πρέπει να μειωθεί. Η χρήση αυτών των χημικών για την καλλιέργεια σόδιων σε ανοιχτούς ε, χώρους της υπαίθρου είναι κάτι που δεν είναι βιώσιμο. Σχεδιασμός των παρασιτοκτόνων είναι δραστικές ουσίες βιολογικά και είναι τοξικές για ζωντανούς οργανισμούς που θεωρούνται ε, παράσιτα για κάποιες καλλιέργειες. Αλλά είναι τοξικές και για άλλους ε, ε, οργανισμούς. Τα πουλιά, τα μικρά θηλαστικά, οι μέλισσες, οι βάτραχοι κλπ. Αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους και για τα ε, ζώα, τα ε, οικόστητα Χιλιάδες όμως τόνοι από αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται και κινδυνεύει το περιβάλλον με αυτόν τον τρόπο και η υγεία. Έχουμε δει ότι επηρεάζεται ο μεταβολισμός, υπάρχει καρκινογένεση, ε, προβλήματα στους καλλιεργητές και στις οικογένειες των καλλιεργητών. Επηρεάζεται και το περιβάλλον. Σε 42% των ποταμιών και των λιμνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οικοσυστήματα υποφέρουν από χρόνια τοξικότητα. Όπως βλέπετε στο χάρτη, οι γκρίζες αυτές ε, σε αγγλικές περιοχές βλέπετε ότι ε, έχουμε πάνω από 75% τοξικότητα και το υπόλοιπο οικοσύστημα ε, απειλείται. Μια μελέτη πρόσφατα απόδειξε ότι έχει, τα, τα, έντομα έχουν μειωθεί κατά 70% στα δάση στη Γερμανία μέσω εντατικής καλλιέργειας και χρήσεως μεγάλης των παρασιτοκτόνων. Τα παρασιτοκτόνα έχουν και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, αρνητικό αντίκτυπο στη γεωργία. Καταστρέφουν ε, το οικοσύστημα, τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, όπως η βιπικιλότητα των εδαφών, η γονιμότητα. Ε, επίσης, γίνονται πια δύναμα τα φυτά, αντιστέκονται τα παράσιτα περισσότερο και αναγκάζονται σε φαύλο κύκλο οι καλλιεργητές να χρησιμοποιούν πιο ισχυρά παρασιτοκτόνο. Πρέπει να τεθεί τέρμα σε αυτή την πρακτική. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο από το αίτημα πέρα από τον κανονισμό για τα πασιτοκτόνα, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησαν οδηγία για τη βιώσιμη χρήση των παρασιτοκτόνων και καλούνται τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τα χημικά παρασιτοκτόνα σαν ίστατη λύση και θα πρέπει να τεθούν στόχοι για τη μείωση τη χρήση των παρασιτοκτόνων. Ολοκληρωμένη διαχείριση αυτών των ουσιών που διαχειρίζεται και δεν εξαλείφει τα παράσιτα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει προληπτικές μεθόδους άμυψη φορά, πολλαπλές οδιές, ε, διάφορα είδη καλλιεργιών, βιολογικές μεθόδους και όταν όλες οι λύσεις αποτύχουν, τότε να χρησιμοποιούνται τα παρασιτοκτόνα. Και τα φυσικά παρασιτοκτόνα συμπεριλαμβάνονται. Όμως, πρόσφατη έκθεση έδειξε ότι οδηγία δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έξι κράτη-μέλη έχουν θέσει σαφείς στόχου μειώσεως παρόλο που υπάρχουν εναλλακτικέ ε, λύσεις. Για να ενστερνιστούν τις εναλλακτικέ, υποχρεωτικοί στόχοι θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα παρασιτοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν ήδη εναλλακτικέ μέθοδοι. Και όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να απαγορεύσουν τη χρήση παρασιτοκτόνων σε δημόσιου πράσινου χώρου. Ειδικά μέτρα θα πρέπει να βάλουν την προστασία των ποταμών και των λιμνών και των διαφόρων οικοσυστημάτων. Μακροπρόθεσμη μείωση μέσω στόχων είναι απαραίτητη για την έγκριση και οθέτηση εναλλακτικών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να βοηθήσουμε τους γεωργούς να κάνουν τη μετάβαση. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά εκπαιδεύοντάς τους, δίνοντάς τους συμβουλές για εναλλακτικέ μεθόδους, για συγκεκριμένες σοδιές και καλλιέργειες. Έρευνα και ανάπτυξη θα πρέπει να εστιάζεται επί εναλλακτικών λύσεων. Η καταστροφή της βιοπικιλότητας όσον αφορά τα αγροκτήματα και τον περιβάλλοντα χώρα. Για να παραχθεί μια σοδιά οικονομικά ενδιαφέρουσα δεν είναι καθόλου βιώσιμο σύστημα και είναι πρόδρομος προς αδίέξοδο. Όσο πιο γρήγορα αλλάξουμε τις πρακτικές, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και το μέλλον των φυσικών μας πόρων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλοι Πρόεδρος. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιθυμούν να σχολιάσουν και πολλές ερωτήσεις. Η κυρία Γκαρντίνη είναι η πρώτη που θέλει τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι όλα είναι καλά και άγια και όλοι συμφωνούμε επί της αρχής, επί των αρχών. Ακούγοντας να αναφέρεται η Γεωργία με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι σκεφτόμαστε μια Γεωργία που δεν υπάρχει πια. Γιατί το λέω αυτό. Όταν πάω εγώ σε συναντήσεις που διαγωνώνει ο κόσμος της Γεωργίας, υπάρχει μια πολύ σύγχρονη Γεωργία όπου μιλάνε για γεωργία της ακρίβειας. Υπάρχουν μηχανήματα που κινούνται μόνοι τους, χωρίς να τους ελέγχει ο άνθρωπος, υπάρχουν δορυφόροι, κάθε τεχνολογία που μας λένε πόσο να χρησιμοποιούμε, τι πράγμα, ελάχιστο. Και τα παρασιτοκτόνα ακριβώς είναι αυτό που θέλαμε, είναι η τελευταία λύση. Όταν υπάρχουν ασθένειες, όταν υπάρχουν βακτηρίδια, όταν υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν τη χρήση του. Πάντα χρησιμοποιούνται όταν πρέπει, εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, στο ελάχιστο δυνατόν με τα αποτελεσματικότερα προϊόντα. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με το πλαίσιο της γεωργίας που παρουσιάζεται σαν μια γεωργία του λίθινης εποχής. Ίσως κάποια συνάντηση περισσότερο, κάποια επίσκεψη παραπάνω στις γεωργικές επιχειρήσεις θα μας οδηγούσε να υφορθώσουμε μια εικόνα ποιος πιο σωστή, τη σύγχρονη γεωργία. Αυτή η γεωργία περιγράφεται εδώ δεν υπάρχει πια, τούτου λεχθέντο. Και εμεί παίρνουμε φάρμακα για να θεραπευτούμε όταν στενούμε. Το ίδιο ισχύει και για τα φυτά. Τα φυτά αρρωσταίνουν και όταν αρρωσταίνουν χρειάζεται φάρμακα, όπω η ξυλέλα φαστιντιόζα. Η ξυλέλα φαστιντιόζα είναι ένα βακτηρίο που δεν, είναι, ε, που δεν θεραπεύεται, είναι ανίατο. Και μπορεί με αυτά τα προϊόντα κάπω να ελεγχθεί. Που μπλοκάρουν του φορεί πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Δεν μπορούμε να θέτουμε αυθαίρετους στόχους. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι καρπός ισορροπίας. Εντάξει, καλό είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ελέγχουν. Πάντα είναι καλό το κίνητρο. Μετά θα πρέπει να καταλάβουν και εκείνοι ότι πρέπει να υπάρξει σωστή ισορροπία. Εκείνοι είναι καλοί θεματοφύλακε υπουργοί. Πρέπει να έχουν στόχου. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Και ρωτώ, όταν λέτε λοιπόν ότι πρέπει να βρεθούν άλλα πράγματα, τι γεωργία θέλετε. Ποια ευρωπαϊκή γεωργία. Έχουμε στόχους, τους πιο αυστηρούς όλων στον κόσμο. Έχουμε, ένα, έχουμε πάρα πολλούς κανόνες να λέτε ότι πρέπει να αλλάξει ο κόσμος της γεωργίας. Πώς ασκούμε τη γεωργία. Ποια έχετε υπόψη σας. Μήπως αυτή για τους πλούσιους, για την ελίτ. Δηλαδή θα πρέπει λοιπόν ή θα πρέπει να απευθύνεται ο, ο κατανοτής προς προϊόντα τον οποίον την προέλευση δεν γνωρίζει. Ευχαριστώ. Κύριε Γκούτελαντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε είναι ένα πολύ ισχυρό, ηχηρό μήνυμα του πολίτε αυτή η πρωτοβουλία. Μόνο τα ασφαλή προϊόντα πρέπει να επιτρέπονται. Αν υπάρχουν επιστημονικέ αμφιβολίες ό,τι αφορά τι επιπτώσει κάποιων προϊόντων, κάποιων ουσιών για το περιβάλλον ή για την ανθρώπινη υγεία, δεν είναι υπεύθυνο από τη δική μα πλευρά απλά αυτομάτω να ε, ανανεώνουμε τι άδειε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση της γλυφωσάτης και είναι κάτι που υπογραμμίζει και ένα δομικό πρόβλημα. Η Ευρώπη δεν κάνει αρκετά για να προωθήσει την ανάπτυξη πιο βιώσιμων εναλλακτικών. Και αυτό είναι εις βάρος και της βιοπικιλότητας αλλά και της ανθρώπινης υγείας. Και έχω και κάποια ερωτήματα για σας ε, κύριε Επίτροπε. Πρώτον, γνωρίζουμε ότι πολλοί γεωργοί χρησιμοποιούν ε, ε, παραστοκτόνα προληπτικά, αντί να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν άλλες εναλλακτικέ. Δεν φταίνει οι γεωργοί. Οι γεωργοί ανησυχούν κυρίω για τη σοδιά τους. Είναι όμως πρόβλημα αυτό για το περιβάλλον και μπορεί επίσης να επιφέρει ε, αρνητικές επιπτώσεις και για τους γεωργούς ε, και την υγεία τους αλλά και τους καταναλωτές. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε εδώ τα κίνητρα ε, και θα ήθελα να ξέρω τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, ήδη κάποια κράτη-μέλη έχουν πάρει κάποια μέτρα για την απαγόρευση της χρήσης ε, ζημιογόνων, ζησανιοκτώνων σε επικίνδυνες περιοχές, σε σχολεία, σε πάρκα, σε παιδικές χαρές, σε φυσικά ε, θέρετρα. Είναι χώρες λοιπόν που είναι διευθυμένες να κάνουν περισσότερα για την προστασία των πολιτών. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Αυτό ζητάμε. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν παίρνουν τέτοια μέτρα. Και νομίζω ότι Πραγματικά εδώ χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή λύση. Και δεν θέλω να ξέρω τι σκοπεύει ε, να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί καθυστερεί, γιατί δεν προτείνει ε, τέτοιου είδου υποχρεώσει να είναι υποχρεωτικέ, ε, τέτοιου είδου απαγορεύσει να είναι υποχρεωτικέ στα κράτη-μέλη. Η ίδια η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βιώσιμη χρήση των ζενιοκτώνων και η σχετική οδηγία δείχνει ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη έχουν μείνει πίσω ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Υπάρχουν μεγάλα κενά στα, στα εθνικά σχέδια δράσης όταν αυτά υπάρχουν. Και αυτή η οδηγία έπρεπε να έχει εφαρμοστεί ήδη το 2012. Έχουμε φτάσει το 2017 τώρα. Αυτή η έκθεση της ε, Επιτροπής για την εφαρμογή λέει ότι η Κομισιόν σκέφτεται να ακολουθήσει τη διαδικασία παραβάση. Ε, τι ακριβώς μπορούμε να δεχτούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάκιντάιρ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ λαμβάνω όλο και περισσότερες επιστολές από ψηφοφόρους γεωργούς που μου λένε, παράδειγμα χάρη, ε, είμαι πραγματικά ιδιασμένη πως ε, τα, τα, πολι, τα επιστημονικά αποτελέσματα ε, παραποιούνται ε, σε, για πολιτικούς λόγους πρέπει επιτέλους να πούμε στο κοινό και να πούμε στους, ε, ε, στο κοινό και στους πολιτικούς συνένοντες ότι η γλυφοσάτη είναι ασφαλή εδώ και 40 χρόνια. Υπάρχουν εκατοντάδες μελέτες που το αποδεικνύουν αυτό. Νωρίτερα αυτό το μήνα άλλη μια ανεξάρτητη μελέτη μακροπρόθεσμη του Εθνικού Ινστιτούτου για τον Καρκίνο δεν βρήκε καμία σχέση μεταξύ της γλυφοσάτης ε, και των λυμφωμάτων των καρκινικών. Εδώ έχω ένα πρόβλημα με το θέμα αυτό. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να μιλάμε για στόχους οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί. Εγώ είμαι υπέρ των στόχων. Και δεν ξέρω κανένα γεωργό που θέλει ε, να εκτίθεται στα χημικά περισσότερα από ό,τι χρειάζεται. Έτσι λοιπόν οι στόχοι που πρέπει να υποστηρίζουμε είναι ε, για την έρευνα για πιο αποτελεσματικές και καλύτερες μεθόδους γεωργίας. Μοντέρνα πολιτική ε, συντήρησης του εδάφους, παραδείγματο χάρη. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια χρησιμοποιώντα ε, ε, φυσικές ε, μεθόδους προστασία του έδαφους από την ε, επιδείνωσή του αλλά χωρίς τη, γλυφο, θα πρέπει να έχουμε πλέον μηχανικό έλεγχο από τους γεωργούς 25% αύξηση της ε, εκπομπής ε, αερίων θερμοκηπίου. Αυτό θα έχει επιπτώσεις ε, για την χλωρίδα, την πανίδα. Πραγματικά θα ήθελα αυτοί που ζητούν πλήρη απαγόρευση να το εξετάσουν το θέμα πιο λογικά, να δουν τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε εδώ. Θέλουμε καλύτερη συντήρηση του εδάφους, θέλουμε καλύτερες μεθόδους γεωργικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ως Γκεμπράντη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τους ε, ανθρώπους που ανέλαβαν αυτήν την πρωτοβουλία των πολιτών. Νομίζω ότι αξίζει να το τονίσουμε αυτό. Και σήμερα βλέπω για άλλη μια φορά πόσο πολλωμένη και συναισθηματικά φορτισμένη είναι αυτή η συζήτηση. Από τη μία η κατάργηση της γλυφοσάτης είναι το τέλος της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων και για τους άλλους η συνέχιση της χρήσης της γλυφοσάτης είναι το τέλος του κόσμου. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές γνωρίζουν πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία τελικά. Αυτό όμως που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι όλο και περισσότερα προβλήματα υπάρχουν λόγω της υπερβολικής χρήσης παρασιτοκτόνων, όχι μόνο της γλυφοσάτης, στη γεωργία μας. 400 εκατομμύρια κιλά ε, παρασιτοκτόνων, μόλις το είδα στη διαφάνεια, είναι τεράστια ποσότητα η μισή γεωργική γη έχει ήδη κορεστεί από τη γλυφοσάτη. Αν δείτε λοιπόν τις μελέτες για τα έντομα και όλα αυτά τα στοιχεία, πραγματικά θα ανησυχήσετε. Για μένα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε φτάσει στα όρια του τρέχοντος συστήματος. Δεν έχουμε εξετάσει επαρκώς ε, τις σορευτικές επιπτώσεις της χρήσης των παρασιτοκτόνων. Δείτε τα ένα-ένα είτε είναι καρκινογόνο είτε όχι, εδώ γι' αυτό μιλάμε, ε, τα σορευτικά, οι σορευτικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στο περιβάλλον είναι τεράστια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια ευρύτερη προσέγγιση και από την πλευρά της Κομισιόν και της ΕΦΣΑ. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως η γεωργία χωρίς χημικά θα είναι ωφέλιμη για όλους μας. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα πρέπει να καταργήσουμε τη γλυφοσάτη. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να πάμε σε μια γεωργία στην Ευρώπη η οποία θα ζει χωρίς τα χημικά. Η μετά των χημικών εποχή. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να μην θέσουμε σε κίνδυνο την γεωργική παραγωγή, αλλά να έχουμε τεράστια ωφέλη για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Ίσως θα πρέπει η Κομισιόν να το δει και αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λίνς, ευχαριστώ. Να επανέλθω στα όσα ακούσαμε στην αρχή αυτού του πάνελ. Νομίζω ότι γενικεύουμε πολύ και δεν περιγράφουμε τα προβλήματα επαρχώς δίνοντας απλές ερωτήσεις. Ε, γενικά ε, κατηγορούμε την εντατική γεωργία και τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα που έχουμε μπροστά στα μάτια μας και το ζητώ. Για παράδειγμα, η γλυφοσάτη χρησιμοποιείται ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι μόνο στη Γεωργία, Ε, ακόμα και, στις, ε, και στην, ε, στους σιδηροδρόμους χρησιμοποιείται, ας πούμε, στη δική μου ε, περιοχή. Καθαρίζουμε τις γραμμές ή ε, χρησιμοποιείται στα παιχνίδια, γενικά στην ιδιωτική ζωή, χωρίς να υπάρχει εμπεριστατωμένη απόδειξη σχετικά με το κατά πόσο είναι βλαβερή ή όχι. Θα έπρεπε λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο περισσότερο αυτά τα θέματα όπως τα παιδικά παιχνίδια, ε, να δούμε κατά πόσο ε, μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση της ε, ή και να την απαγορεύσουμε. Ας πούμε, στη δική μου πατρίδα πέρυσι δόθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε παρασιτοκτόνα από ό,τι στο παρελθόν. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για μείωση και αυτό ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριο Δήμες Μέκερ. Ευχαριστώ πολύ. Καλω ορίζω όλους όσους συμμετέχουν στη συζήτηση. Πολλοί πολίτες ανησυχούν για το θέμα αυτό, για τη χρήση των ε, παρασιτοκτόνων είναι μεγάλη πρόκληση η μείωση της χρήσης αυτών των ουσιών και να εγκαταλειφθούν οι δυνατόν και να έχουμε τύχει στο τέλος. Θα πρέπει ε, να χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο. Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς να υπάρχει ανάγκη, πιστεύω, αυτές οι ουσίες. Υποστήριξα το στόχο που εκφράστηκε για τη γλυφοσάτη, αλλά ας δούμε τη γενικότερη εικόνα. Έχουμε την έκθεση της 10 Οκτωβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχέδια δράση των κρατών μελών και την πρόοδο όσον αφορά τη βιώσιμη χρήση των παρασιτοκτόνων. Εκεί θα δείτε ότι πόρο απέχουμε από τους στόχους. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Παραδείγματο χάρη, από ό,τι φαίνεται, η ολοκληρωμένο, ολοκληρωμένος έλεγχος των παρασίτων δεν χρησιμοποιείται παρκώς και τα κράτη-μέλη δεν πετυχαίνουν τους ποσοτικούς τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα στους διάφορους τομείς δράσης, προτείνεται δεσμευτικούς στόχους μειώσεως όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάζοντας αυτή την πρόταση, εγώ τι λέω. Χρειαζόμαστε η καλύτερη εφαρμογή καταρχήν της ισχύουσας οδηγίας στα κράτη-μέλη. Και αυστηρότερη εφαρμογή και έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων. Θα πρέπει ο στόχος της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρασίτων χρησιμοποιείται επαρκώς. Σε αυτό το πλαίσιο, πώς θεωρείτε, ποια είναι η άποψη για την έξι Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη χρήση των παρασιτοκτόνων, τι προοπτικές υπάρχουν για τη μέγιστη χρήση των υπαρχόντων εργαλείων, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση. Η άποψή σας για τη νέα ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποια είναι, για την ανταλλαγή πληροφοριών για βιώσιμη χρήση των παρασιτοκτόνων είναι πιο εύκολη η πληροφόρηση των ε, πολιτών με αυτόν τον τρόπο. Να προσθέσω ότι όσον αφορά τη Φλάνδρα στη χώρα μου, από το 2015 είχαμε απαγόρευση των παρασιτοκτόνων από πλευρά τη τοπική αυτοδιοίκηση. Λέμε ότι χωρί είναι πιο υγιεινά τα προϊόντα, χωρί παρασιτοκτόνα. Αυτή είναι μια δράση που πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω, με τα χαρά να ακούσω αν συμφωνείτε μαζί μου ή όχι. Τέλο, βέβαια, ένα θέμα που συνδέεται με τη γεωργική πολιτική. Πιστεύετε κι εσείς ότι είναι σωστή προσέγγιση. Ο κ. Μαρτελέζη έχει το λόγο. Eh, Να ευχαριστώ καταρχήν όλους όσους πήραν την πρωτοβουλία αυτή, την πρωτοβουλία πολιτών και βεβαίως και όσους υπέγραψαν το 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία, με βάση την αρχή τη προφύλαξη, αλλά και με βάση το σκάνδαλο μετά τα, τα έγγραφα του Μονσάντο, συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση να καταργηθεί η γλυφοσάτη. Να πω ότι οι πράσινοι Ευρωπαίοι, επειδή υπάρχει έλλειψη διαφάνεια τη ΕΦΣΑ, έχουμε στείλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την ε, έλλειψη πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα. Μιλάμε για προ, προσωρινή, ε, σταδιακή κατάργηση τη γλυφοσάτη, όπω λέει το Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βρούμε και εναλλακτικέ. Και όταν μιλάμε για εναλλακτικέ, εννοούμε εναλλακτικέ που θα διαφυλάσσουν την υγεία των πολιτών, τη βιοπικιλότητα, το έδαφο αλλά και τα ζώα. Εδώ δεν μιλάμε για ένα προϊόν, μιλάμε για ένα μοντέλο. Ένα μοντέλο που αυτή τη στιγμή είναι τοξικό για του ανθρώπου για το περιβάλλον. Χρειάζεται λοιπόν μία εξέλιξη από το αγροβιομηχανικό μοντέλο σε ένα μοντέλο αγροοικολογικό που να μην δουλεύει σε βάρος της φύσης αλλά υπέρ της φύσης. Μιλάμε για νέες τεχνικές, μηχανικές, βιολογικές ε, ε, και βεβαίως μιλάμε και για μια ε, αγροτική οικολογία που θα καταρτίζει τους γεωργούς, τους εργαζομένους, θα ανταλλάζουν εμπειρίες, γνώσεις μεταξύ τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πολιτική που να είναι συνεπής με τις πολιτικές βιοπικιλότητες και με τις πολιτικές που αφορούν την, αλλαγή, την κλιματική αλλαγή. Εξού και το πολύ σημαντικό θέμα της προφύλαξης, της διαφύλαξης του εδάφους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κύριε Επίτροπε, στα μέσα που έχουμε στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής για τη χρηματοδότηση αυτής της μετάβασης, να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα αυτά. Το πυλώνα τη γεωργική ανάπτυξη, παραδείγματο χάρη. Κύριε Επίτροπε, επίση πρέπει η Κομισιόν με πιο αποφασιστικό τρόπο να στηρίξει ένα αγροβιολογικό μοντέλο. Θέλω να ξέρω τι πιστεύει η Κομισιόν γι' αυτό. Αντί για ένα μοντέλο αγροβιομηχανικό, να ε, προκρίνουμε ένα μοντέλο αγροβιολογικό. Και βεβαίως να, να ρωτήσω και, τους, και την πρωτοβουλία των πολιτών αν και αυτοί υποστηρίζουν ένα τέτοιο μοντέλο. Ευχαριστώ. Κύριος Ευχαριστώ. Ε, πρέπει να μιλήσουμε, αυτό είναι η επικεφαλίδα, γιατί κανείς ε, δεν κατανοεί την κοινωνία και δεν μιλάμε και ανοιχτά. Δεν υπάρχουν ριζικές ε, λύσεις. Η φύση δίνει κάποιες λύσεις σε μία γεωργία χωρίς χημικά θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε την οργανική την ανόργανη χημία. Η ανόργανη χημία επίσης ε, προσωμιάζει τις διαδικασίες των, των οργανικών ενώσεων και γενικά φαίνεται πως ε, ε, δεν μπορεί να υπάρχει γεωργία χωρίς χημικά. Τώρα, ερώτημα. Ε, αν θέλουμε αυτή, αυτός ο περιορισμός ε, στο χρόνο να γίνει τελικά κατάργηση, ε, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος τελικά. Δεύτερον, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, κύριε Επίτροπε, ποιον θα ωφελήσει αυτή η ευρωπαϊκή απαγόρευση, ίσως τον ανταγωνισμό και τρίτον για, την, για το κίνημα των πολιτών. Δεν θα έπρεπε να ασχοληθείτε το ίδιο και με την ε, γενετική τεχνική, ε, όπως κάνετε και με τα χημικά, γιατί τι θα γίνει αν χρησιμοποιείτε και αυτή. Θα πρέπει λοιπόν για την αξιολόγηση των κινδύνων να πούμε ότι ε, αν διαπιστώσουμε ότι η γλυφοσάτη είναι καρκινογόνος, ε, η οποία βρίσκεται στο κρέας, ε, στα αναβολικά παντού, ε, θα πρέπει να απαγορευτεί και θα πρέπει να βρούμε και τα μέσα για να το κάνουμε. Mr. Ο κύριος Χάουσλινγκ. Ε, η γενετική τεχνική οδηγεί σε περισσότερη χημεία. Το ίδιο γίνεται και στην Αμερική με τη γλυφοσάτη, το ίδιο και στη Γερμανία. Η γενετική τεχνολογία λοιπόν δεν είναι εναλλακτική. Ε, μιλάμε για τη γλυφοσάτη, μεγαλόφωνα και τα λοιπά, να είμαστε ειλικρινείς. Αν μιλήσουμε με τους γεωργούς, η γλυφοσάτη ε, είναι... Ε, φθηνή, τη χρησιμοποιούν και βρά γρήγορα, τους εξοικονομεί εκατοντάδες ευρώ. Ε, δεν μπορούμε πια να την σκεφτούμε τη γεωργία χωρίς ε, τη γλυφοσάτη. Ε, καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν στη γεωργία πλέον και δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτά παρόλο που βλάπουν τον το περιβάλλον. Η χημεία στην γεωργία ε, έχει κάποια χρήση και καλό θα ήταν μεν να ε, υπάρχει μια μείωση αλλά όχι τελείως κατάργηση. Επίσης ε, θα πρέπει να πούμε στην Κομισιόν ότι η γλυφοσάτη ε, μέσα από σύγχρονες μεθόδους εναλλακτικές θα μπορούσε να αντικατασταθεί. Γιατί αγνοεί λοιπόν η Κομισιόν αυτή την απώλεια της βιοποικιλότητας, δεν το καταλαβαίνω. Το 80% των εντόμων χάνονται. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τη γεωργία και τη χημεία. Φυσικά και έχει να κάνει. Πρέπει να κάνουμε ειλικρινή συζήτηση. Και μετά τίθεται και το ερώτημα στην Κομισιόν και ίσως και στην Πρωτοβουλία ε, κατά πόσο η Κομισιόν και η Ευρώπη εκβιάζονται όταν υπάρχουν ε, ε, απειλές ε, για μηνύσεις από την πλευρά των παραγωγών της γλυφωσάτης. Εμείς θέλουμε μια συγκεκριμένη μορφή γεωργίας και δεν θα εκβιαστούμε από τις επιχειρήσεις. Αυτό θα πρέπει να πει η Κομισιόν. Εδώ ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Λύση Μάχου έχει το λόγο τώρα για ένα τέταρτο για να μπορέσει να απαντήσει στα υποθέντα. Um, it's very sad to see. Είναι θλιβερό που βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν λάβει στα σοβαρά ε, την οδηγία για τη βιώσιμη χρήση αυτών των ουσιών. Γι' αυτό προτείνουμε υποχρεωτικούς στόχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε ότι μόνο πέντε κράτη-μέλη στα σχέδια δράσεώς τους έχουν συγκεκριμένους προσμετήσιμους στόχους και λένε ότι θα πετύχουν αυτούς τους στόχους. Θέλουμε να το κάνουν και τα 28 κράτη-μέλη και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παίξει ένα ρόλο σε αυτό. Σχετικά με αυτά που υπόθηκαν για τη Γεωργία από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Υποστηρίζουμε 100% την σωστή Γεωργία δεν μπορούν ξαφνικά όλοι οι γεωργοί να αλλάξουν μεθόδους και να χρησιμοποιήσουν, ε, να έχουν βιολογικές καλλιέργειες, αλλά υπάρχουν εργαλεία να τους βοηθήσουμε να κάνουν τη μετάβαση. Δεν μιλάμε για θαύματα, αλλά είναι κάτι εφικτό. Πρέπει πολλές τεχνικές και μέθοδοι να χρησιμοποιηθούν, ούτως ώστε να συμβεί αυτό που θέλουμε και να υπάρχει και η προθυμία των καλλιεργητών να το κάνουν. Αυτό, καθώς και οι πολιτικοί πρέπει να έχουν την ίδια βούληση είναι μια απόφαση που θα πρέπει σε κάποιο σημείο να ληφθεί. Σήμερα ή όταν τα οικοσυστήματά μας ε, απειλούνται ακόμα περισσότερο από ό,τι τώρα. Δεν παρουσίασα όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε για την επιδείνωση του περιβάλλοντος λόγω παρασιτοκτόνων. Αληθεύει ότι η μελέτη των γερμανικών δασών αναφέρει την εντατική γεωργία και τη χρήση των παρασιτοκτόνων μαζί με την αλλαγή του κλίματος έχουν προσμετρήσιμα στοιχεία όσον αφορά τα κατάλοιπα παρασιτοκτόνων στο νερό. Οι τιμέ, από ό,τι θυμάμαι, είναι από 85 μέχρι 91% ε, το πρόβλημα οφείλεται στα παρασιτοκτόνα όσον αφορά τα κατάλοιπα στο νερό. Οι τρόποι χρήσεως επηρεάζουν την ύπαρξη των καταλήπων στα ύδατα εμείς υποτιμούμε την τοξικότητα που παράγουμε μέσω της χρήσης προσιτοκτόνων στο περιβάλλον και στα ύδατα. Και δεν αφορά μόνο την οδηγία τη βιώσιμη χρήση. Έχουμε και την οδηγία πλαίσιο για το νερό, για το πόσιμο νερό επίσης την άλλη οδηγία. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, υφίσταται, πρέπει να εφαρμοστεί. Να είμαστε σίγουροι ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να μιλήσουμε στους γεωργούς. Να τους ρωτήσουμε, μπορούν να ζήσουν χωρίς τη γλυφοσάτη. Υπάρχουν πολλοί γεωργοί που δεν χρησιμοποιούν τη γλυφοσάτη. Καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι δύσκολο να αλλάξουν οι άλλοι γεωργοί. Έχουν πολλές, πολλές καλλιέργειες, χρησιμοποιούν πολλές εναλλακτικέ μεθόδους οι γεωργοί Κάποιοι έκαναν τη μετάβαση, ε, ήταν δύσκολο, αλλά τα κατάφεραν. Οι άλλοι γεωργοί δεν μπορούν να το κάνουν. Αν έχεις 2.000 εκτάρια με στάρι, δεν μπορεί να το κάνεις, με δημητριακά. Αν έχεις 2.000 εκτάρια με 5 ή 6 καλλιέργειες και δημιουργείς αμυψισπορά και άλλες μεθόδους που υπάρχουν, μπορείς να το καταφέρεις. Να χρησιμοποιήσεις και την τεχνολογία. Δεν θα σωθεί το μέλλον της γεωργίας μέσω ξηρασία και μέσω χρήσεως ε, των παρασυτοκτόνων στι εκμεταλλεύσει. Μπορούμε να έχουμε καλύτερη τεχνολογία, να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα GPS, μπορούμε να ελέγχουμε την υγρασία, τα παράσιτα, να βρούμε πότε εμφανίζονται αυτά και μπορούμε να συνεργαστούμε με τα παράσιτα. Ίσως να μην είναι όλα κακά. Ε, ίσως δεν χρειάζεται να απελευθερώνουμε όλα αυτά τα χημικά στο περιβάλλον και θα είναι και φθηνότερη μια άλλη λύση. ίσως δημιουργήσουμε μεγαλύτερη απασχόληση, γίνει και άλλη έρευνα. Και τελικά θα καταλήξουμε σε ένα μέλλον που δεν θα χρησιμοποιούμε τα παρασιτοκτόνα. τις σημειώσεις μου τώρα για τη βιώσιμη χρήση των παρασυντοκτώνων και τη σχετική οδηγία. Γιατί δεν την εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη, γιατί δεν εφαρμόζουν την προστασία των ε, συστημάτων, των υδατικών συστημάτων. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά παρασιτοκτόνα, παρά κατάλοιπα από παρασιτοκτόνα στα ύδατα. Σε κάποιες χώρες έχουν κάποιες ζώνες προστασίας, ε, απομόνωσης και άλλες δεν έχουν διαχωριστικές περιοχές. Πώς θα τα καταφέρουμε αν δεν τηρούνται οι στόχοι και αν δεν γίνεται σεβαστή οδηγία. Μειούμε για στόχους, μείωση η Γαλλία είπε ότι 25% θα είναι η μείωση μέχρι το 2020 και 50% μείωση των παρασιτοκτόνων μέχρι το 2025. Γιατί δεν παρενούμε και άλλες χώρες να κάνουν κάτι παρόμοιο, όπως η Γαλλία. Η μόνη επιτυχής προσέγγιση και υλοποίηση οδηγία είναι ότι σταματήσαμε, φαίνεται, τους αεροψεκασμούς, παρόλο που χρησιμοποιείται αεροψεκασμοί με κάποιες παρεκκλήσεις. δείτε αυτό μια επιτυχία που δεν γίνονται αεροψεκασμοί πλέον οι άλλε αρχέ για τη βιώσιμη χρήση των παρασυντοκτώνων και τη σχετική οδηγία. Πώ θα εφαρμοστούν οι άλλε αρχέ. Ο Επίτροπο τι πιστεύει. Πώ θα προχωρήσουμε χωρί άλλη πίεση να πετύχουμε του στόχου. Τα κράτη-μέλη το 2018 πρέπει να υποβάλουν στόχους. Παραμένουν 23 κράτη-μέλη Ίσως πρέπει να είναι πιο αυστηροί στόχοι. Ίσως πρέπει να ακολουθηθούν κάποια παραδείγματα. Φοβούμαι ότι, ότι οι υπόλοιπες ερωτήσεις αφορούσαν εσάς κύριε Επίτροπε. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Πάολα Κολόμπα, υπεύθυνη για ελέγχους και αναλύσεις στον τομέα της υγείας. Έχετε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως, όπως ε, έχουν ήδη πει πολλοί, αλλά και οργανωτές ε, της πρωτοβουλίας, η βιώσιμη χρήση των Ζανιοκτών και σχετική οδηγία είναι εξαιρετικά κρίσιμο εργαλείο για τη μείωση του κινδύνου για την υγεία και το περιβάλλον από τα ζανιοκτώνα. Και αυτό το εργαλείο είναι στα χέρια των κρατών μελών. Τους έχει ζητηθεί από την οδηγία να περιγράψουν στα εθνικά τους σχέδια δράσης πώς σκοπεύουν να ε, ανταποκριθούν σε αυτά που προβλέπει αυτή η οδηγία και πρέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης να, προβλέπει, να προβλέπει ποσοτικούς στόχους ε, μετρήσιμους και χρονοδιάγραμμα. Ξέρετε ότι η Κομισιόν πρόσφατα ανέκρινε μία έκθεση. Μία έκθεση που δεν βασίζεται μόνο στην ανάλυση των, των σχεδίων δράσης, αλλά και στις δικές μας διαδικασίες ελέγχου. Έχουμε λοιπόν μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει σε επίπεδο κρατών μελών. Όχι μόνο ε, δηλαδή με βάση τις, αυτά, τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Ε, είναι γνωστό ότι η Κομισιόν δεν είναι και τόσο ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα των κρατών μελών. έχει χαθεί μια ευκαιρία έως τώρα, το λέμε και στην έκθεση και το λέμε και σε κάθε κράτος μέλος ε, ε, επιμέρους. Τους λέμε δηλαδή τι λείπει στα δικά τους σχέδια και τι περιμένουμε να δούμε στο μέλλον, στα μελλοντικά σχέδια δράση. Του 2018 δηλαδή. Υπάρχουν δύο κεντρικά ζητήματα όπου θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους. Το πρώτο είναι η έλλειψη στόχων για τη μείωση του κινδύνου. Έχουμε δει πέντε καλά παραδείγματα. μας χάρη η Γαλλία έχει θέσει ένα στόχο για τη μείωση ε, ε το, της χρήσης ανεοκτώνων. Γιατί να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα. Η Δανία επίσης έχει θέσει ένα τέτοιο στόχο, αλλά ε, γρήγορα διαπίστωσε ότι δεν είναι ο καλύτερος δυνατός στόχος αυτός. Το να μιλάμε δηλαδή για τα μεγέθη δεν αρκούν για να αποδείξουμε ότι μειώνεται ο κίνδυνος. Γι' αυτό λοιπόν και η Δανία αλλά και άλλα κράτη-μέλη σιγά σιγά πάνε προς άλλου τύπου στόχους. στόχους. Ένα άλλο ζήτημα όπου δεν είμαστε τόσο ικανοποιημένοι με τα κράτη-μέλη ε, είναι η εφαρμογή της ε, ολοκληρωμένης διαχείρισης ε, ζυζανίων παρασίτων. Ε, πρέπει να πάμε προς μια, μια διαφορετική, πιο βιώσιμη γεωργία και αυτό το εργαλείο υποχρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη. Αυτό που δεν συμβαίνει είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν ελέγχουν τη συμμόρφωση ε, σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτού του ολοκληρωμένου, διαχείριση. Είναι ένα εργαλείο όπου τα κράτη-μέλη θα πρέπει πραγματικά να ενισχύσουν τι προσπάθειές τους. Ε, τώρα είναι κάποια σχόλια που αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να βελτιώσει την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Πρώτα απ' όλα, όπως ελέγχθη, θα αξιολογήσουμε τα εθνικά σχέδια δράσης, θα δούμε αν τα κενά τα οποία έχουμε εντοπίσει ε, θα ε, καλυφθούν και θα συνεχίσουμε βεβαίως τη δραστηριότητα ε, εποπτείας, παρακολούθησης. Αρχίζουμε τώρα, κατά όλη τη διάρκεια του 2018, ελέγχους για να ελέγξουμε, για να επαληθεύσουμε τη συμμόρφωση των κρατών μελών με αυτά που προβλέπει αυτή η οδηγία. Επίσης ε, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη και τα υποστηρίζουμε με την ανταλλαγή βαλίστων πρακτικών. Ε, υπάρχει μια νέα ιστοσελίδα που είναι αρκετά πλήρης ε, σε σχέση με το τι κάνουν τα κράτη-μέλη και την ανταλλαγή βαλίστων πρακτικών. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Έχετε ένα λεπτό, κυρία Λυσιμαχού, εφόσον το επιθυμείτε. Ναι. Λέμε εδώ ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο λειτουργεί ε, ο εξοπλισμός τους ε, ε, έτσι αντιλαμβανόμαστε την οδηγία για τη βιώσιμη χρήση εξετάζουμε κατά πόσο ο εξοπλισμός που ψεκάζει, ψεκάζει λιγότερο περισσότερο και κάτι άλλο που αναφέρθηκε για τα στοιχεία για την παρακολούθηση. Εγώ παρουσίασα κάποια δεδομένα για την τοξικότητα ε, για το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι ο αντίκτυπο αυτών των ζανιοκτώνων ε, στα εδάφη μα. Αναφέρθηκε μια άλλη μελέτη όπου που λέει ότι 45% των εδαφών περιλαμβάνουν γλυφοσάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλα ζανιοκτώνα περιλαμβάνουν. Γνωρίζουμε πόσα βρίσκονται στο νερό, ε, στις λίμνες, στα πάρκα μας. Ε, χρειάζονται περισσότερα στοιχεία λοιπόν και από την τομέα της γεωργίας αλλά και από σε ό,τι αφορά χώρους. Μάλιστα, ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος και τώρα θα περάσουμε στις τελικές δηλώσεις. Κύριε Επίτροπε, κάτσατε μέχρι τώρα, έχετε το λόγο. Πολλά υπόθηκαν, πολλοί απευθύνθηκαν στην Κομισιόν. Ναι, ευχαριστώ. Είναι η καιρός η Κομισιόν να ακούσει εσάς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το ευρύτερο πλαίσιο των διαφόρων ζητημάτων και πραγματικά με μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή άκουσα τις απόψεις και τη συζήτηση που ξεκίνησε μετά από την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών για τη γλυφοσάτη και γενικά για τα παρασιτοκτόνα. Τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το σύστημα διοδότησης και έγκρισης των ζυζανιοκτώνων αλλά και σε σχέση με το πώς ε, γίνονται οι μελέτες αλλά και πώς γίνεται η αξιολόγηση κινδύνων. Εκφράστηκαν ανησυχίες για τη χρήση και τον έλεγχο των παρασιτοκτόνων. Πραγματικά είναι ένα θέμα υψηλής ευαισθησίας, ιδιαίτερα ευαίσθητο ε, και ανακοινεί τα συναισθήματα, πραγματικά ε, πολύ δυνατά συναισθήματα βλέπω και εδώ η Κομισιόν προσπαθεί με κάθε τρόπο να δίνει την κατάλληλη απάντηση στις ε, νομιμοποιημένε νομιμοποιημένες ανησυχίες των πολιτών. Ε, θα λάβουμε υπόψη μας όλα όσα είπατε, ε, θα τα σκεφτούμε και ευχαριστώ και όλους τους συμμετέχοντες για την συνεισφορά τους. Να επαναλάβω την πεποίθησή μου ότι η ενεργός και επικοδομητική δράση μπορεί να συνεισφέρει σε ένα καλύτερο καθορισμό των μελητικών πολιτικών, της κοινή αγροτικής πολιτικής κτλ. Θα ε, σκεφτούμε και θα λάβουμε υπόψη μας όλα τα ζητήματα που τέθηκαν και τις απόψεις που ακούστηκαν. Εμείς απαντήσαμε ε, μέσω του πρόεδρου μας με τη μορφή ανακοίνωσης. Ε, ε, σήμερα έχω πολύ περιορισμένες απαντήσεις γιατί θέλω για άλλη μια φορά να εξετάσω τα ερωτήματα και τα ζητήματα που τέθηκαν. Είναι πρόημο να πω κάτι παραπάνω. θα απαντήσουμε με την τελική μας ανακοίνωση και την προσέγγιση, την τελική της ε, Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Και τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Κρίστοφ Μπάουτς που είναι ε, ε, εκπρόσωπος της Επιτροπής για πέντε λεπτά. Ο κύριος Μπάουτς, ναι, ευχαριστώ. 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν την πρωτοβουλία των πολιτών και σίγουρα όπως ε, φάνηκε από τα όσα μας είπαν, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Ευρώπης υποστηρίζει τα αιτήματά μας να απαγορευτεί η γλυφοσάτη. Εμείς ε, οι πολίτες έχουμε μια κοινή ανησυχία. Υπάρχει αυτή η υποψία που πλανάτε εδώ στην αίθουσα, κατά, όπως ε, κατέδειξε και ο ΠΟΗ, ότι μπορεί η γλυφοσάτη να είναι καρκινογόνος. Υπάρχει ανησυχία ε, για το πόσο μαζικά η γλυφοσάτη βλάπτει μικροοργανισμούς ε, και στο έδαφος και στο πεπτικό σύστημα των εμβιονόντων. Φαίνεται πως η γλυφοσάτη ευθύνεται για το θάνατο των εντόμων και για τις δραματικές αυτές συνέπειες που ακούσαμε και είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες 76% περιορισμός της ε, ε, βιοπικιλότητας ε, των εντόμων στη Γερμανία και αν αυτό το δείτε και σε σύγκριση με τις επιπτώσεις στη γεωργία πραγματικά ε, η αριθμή είναι ακόμα πιο δραματική. Ανησυχούμε λοιπόν ως πολίτες ε, της Ευρώπης και πραγματικά μας εντυπωσιάζει αρνητικά η μαζική επιρροή της Μονσάντο. Ε, και στις διαδικασίες αξιολόγησης και εκτίμησης ε, μέσα από την ΕΦΣΑΤ και την ΕΤΣΑ και μέσα από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Αξιολόγηση των Κινδύνων. Ανησυχούμε επίσης ε, και για αυτό που προέκυψε ότι τελικά τα Μονσάντο papers ακριβώς δείχνουν πώς ε, επέκρυψε ε, η θελημένα η Μονσάντο τους ε, κινδύνους ότι δεν έδειξε τις αντίστοιχες εκθέσεις που και μελέτες που έδειχναν αντίθετα αποτελέσματα και ότι αποκρύψανε κάποιες άλλες μελέτες από εγκεκριμένους επιστήμονες. Επίσης ε, υπάρχει λογοκλοπή. Πραγματικά υπάρχουν ε, τεράστια κομμάτια από τις εκτιμήσεις και τις αξιολογήσεις της Μονσάντο που έχουν περάσει στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματικά τώρα ε, είμαστε αντιμέτωποι και με απειλές από την πλευρά της ε, Μονσάντο ε, για μηνύσεις, για πράγματα για τα οποία ανησυχούν οι πολίτες. Ανησυχούμε, ξανιστάμεθα και πραγματικά είμαστε Ευρωπαίοι, δεν είμαστε απλώς σκεπτικιστές, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ε, και θεωρούμε ότι μόνο όταν δράσουμε μαζικά και ομαδικά θα έχουμε καλύτερη προστασία της υγείας μας, θα ξεπεράσουμε αυτά τα ε, προβλήματα και θα βρούμε τις λύσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν ε, αυτοί, αυτοί οι πολίτες γεμάτοι ελπίδα κοιτούν προς την Ευρώπη, προς τις Βρυξέλλες. Ε, για να δουν τι θα γίνει με την ψηφοφορία για το face out ε, για πέντε χρόνια. Όμως δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Ε, θέλαμε κάτι άλλο. Πάντως και με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και η Κομισιόν. Ο κύριος Ανδροκαίτης πέρυσι τον Ιούλιο σε μια συνέντευξη είπε ότι δεν θέλουν για άλλη μια φορά να διαδοτήσουν τη γλυφοσάτη χωρίς την ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση. Ελπίζω τελικά ε, να μην επηρεαστείτε από τη Μοσάντο και να παραμείνετε πιστός σε αυτό που είπατε τον Ιούλιο. Να μην δοθεί αδειοδότηση στην ε, γλυφοσάτη μέχρι το Δεκέμβρη. Θεωρώ ότι η απόφαση για τη γλυφοσάτη αποτελεί και μήνυμα. Είναι ένα σύμβολο ε, και των φόβων αλλά και των απαιτήσεων των πολιτών της Ευρώπης ε, ε, να ακουστούν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να υπάρξει η απαγόρευση της γλυφοσάτης, αλλά και μία μεταρρύθμιση και αναθεώρηση της διαδικασίας αξιολόγησης των παρασιτοκτόνων αλλά και να υπάρξει μεσοπρόθεσμα μια σταδιακή παρέτηση από τα ε, παρασιτοκτόνα να βρεθούν εναλλακτικές για να μπορέσουν οι πολίτες της Ευρώπης να έχουν και πάλι μια ευκαιρία. Ε, θα ήταν μοιραίο να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και τις επόμενες ημέρες ε, και εβδομάδες να μην ε, στείλουμε αυτό το μήνυμα και να μιλήσουμε ξεκάθαρα για την απαγόρευση της γλυφωσάτης. Σας ευχαριστώ. Να πω μια φράση, λέει ο Επίτροπος. Συγγνώμη κύριε Μπάουτ. Είπατε ότι πιέζεται από τη Μονσάντο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστέψτε με. Όχι. Εγώ δεν είμαι κάποιος που μπορεί να πιεστεί από κάτι κάποιον. Με παρακολουθούσε η KGB, η KGB, ήμουν στη φυλακή, ήμουν κατά του ολοκληρωτικού καθεστώτος Σοβιετικής Ένωσης, η Μονσάντο έχει λιγότερη δύναμη, αφού δεν με πίεσαν αυτοί, δεν με πιέζει η Μονσάντο. Δεύτερον, η υπόσχεσή μου δεν εγκρίθηκε χωρίς ειδική πλειοψηφία δεν κρίνεται χωρίς ειδική πλειοψηφία. Αυτό προσπαθώ. Και ξέρω και εσεί ξέρετε στου Ευρωπαίου ότι το κράτο δικαίου και ότι κυβερνά ο νόμο. Είναι βασικοί κανόνε Κράτο δικαίου και επιβολή του νόμου. Και εγώ θα υπερασπιστώ τελευταία αυτή θέση, να συμμορφωνόμαστε με τον νόμο. Κράτο δικαίου και ότι πρέπει να δικούμε και να κυβερνάμε μέσω του νόμου. Αυτέ είναι οι θέσει μου. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την ακρόαση, ιδιαίτερα τον Επίτροπο τον κύριο Ανδρουκάητη, τα μέλη της Επιτροπής των Πολιτών, ευχαριστώ, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας ευχαριστώ. Τι ακολουθεί, όπως είπε ο κύριος Επίτροπος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιδράσει επισήμως στην πρωτοβουλία αρχές Ιανουαρίου το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις εφόσον έχουμε ενδιαφέρον για το θέμα και δείξαμε ότι είμαστε πρόθυμοι να δραστηριοποιηθούμε για το θέμα λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι πολίτες να εμπιστεύονται τη διαδικασία αξιολογήσεως του κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κυρίως για χρησιμοποιούμε ένα προϊόντα όπως η γλυφοσάτη γι' αυτό Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, εμείς θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Στους, ευχαριστώ τους συμμετέχοντες και καλό σας βράδυ. Και από ερμηνεών. γεια σας, καλό βράδυ.